So good afternoon everybody. Colleagues, please take your seats. We definitely have Συνάδελφοι, καθίστε. Συγγνώμη, ναι, που ξεκινάμε έτσι γρήγορα, αλλά είναι, έχουμε πολλά στην ατζέντα μας σήμερα. Να ξεκινήσουμε με την έγκριση των πρακτικών. Μετά από συμφωνία με τους εισηγητές, το σημείο 5 για τα νέα τρόφιμα και το 6 για τις ε, καλλιέργεια γάματα ομίκρων. έχουν αλλάξει σειρά το ένα μετά άλλο. Αν δεν έχετε αντιρρήσεις, να εγκρίνουμε την ημερήσια διάταξη με την ε, αλλαγή αυτή. Μάλιστα. Και περνάμε τώρα στο δεύτερο σημείο. Ανακοινώσει του Πρόεδρου. Είμαι ιδιαίτερα ευτυχής που καλωσορίζω εδώ α, ε, από το γερμανικό Bundestag, ε, το γερμανικό κοινοβούλιο, μέλη της Επιτροπής Περιβάλλοντος που έχει καλέσει ο Ματία Γκρότε. Έχει καταφτάσει η ομάδα αυτή ή όχι ακόμα? Α, όχι. Ναι, εντάξει, εντάξει, δεν έχει λοιπόν καταφτάσει, δεν του καλωσορίζω κι εγώ ακόμα. Θα τα ξαναπώ μετά. Α, μάλιστα. Κατά δεύτερον, από τις 5 μέχρι τις 7.30 στις 25 Νευρίου θα διοργανώσουμε μια ενημέρωση για το διακυβερνητικό πάνελ για την αλλαγή του κλίματος, IPCC. Ο δόκτωρας Πασάουρη θα κάνει μια κεντρική ομιλία μετά από την επίσημη έγκριση ο, από όλες τις κυβερνήσεις ε, της ε, συνθετικής έκθεσης της ε, πέμπτης συνόδου του IPCC στην Κοπενχάγη και αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον ιδιαίτερος για όσους συμμετέχουν στην COP20 στη Λίμα από πλευρά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά φυσικά και όλα τα μέλη είναι ευπρόσδεκτα. Κάτι άλλο. Η υποστήριξη σχεδίασης ε, για το ODST θα διατεθεί σε τροπολογίες που θέλουν τα μέλη να καταθέσουν για τα νέα τρόφιμα του κυρίου Νίκολσον Το βιστή αποτελεί μια εμπιστευτική υπηρεσία για να σας βοηθήσει όλους στην κατάρτιση τροπολογιών, μια γλωσσική, ένας γλωσσικό έλεγχος, αλλά και πιο συγκεκριμένη βοήθεια. Και έχουμε στείλει ένα σχετικά email από πλευρά της γραμματεία τη Επιτροπής για να ενημερώσουμε τα μέλη. Έχετε διερμηνία σήμερα σε 21 γλώσσες εστονικά και μαλτέζικα δεν έχουμε μόνο σήμερα. Και ως συνήθως έχετε στην διάθεσή σας ε, τα έγγραφα της συνεδρίασης μέσω της εφαρμογής e-meeting και επίσης μεταδίδεται στο διαδίκτυο η συνεδρίασή μας σήμερα. Και από ό,τι φαίνεται θα καταφέρουμε να καλωσορίσουμε τελικά την ομάδα των μελών της Επιτροπής Περιβάλλοντος του Γερμανικού Bundestag. Καλώς ορίσατε και στα γερμανικά, λέει ο Πρόεδρος. Ελπίζω να περάσετε καλά σήμερα στη συνεδρίασή μας. Καλώς ορίσατε. So, uh... Last thing. Τελευταίο σχόλιο σε ό,τι αφορά το 2 της ανακοινώσεις του Προέδρου τα αποτελέσματα της συνεδρίασης των συντονιστών της 25 Σεπτεμβρίου σε ό,τι αφορά τις συστάσεις, τις έχετε λάβει ηλεκτρονικά. Αν δεν έχετε οποιαδήποτε αντίρρηση, θα θεωρηθεί ότι εγκρίνονται. Μάλιστα, έτσι φαίνεται λοιπόν. Για το 3 τώρα το 4 μάλλον διορθώνει ο πρόεδρος της ημερήσιας διάταξης. Σημαντικό ζήτημα. Όπως θα θυμάστε αρισμένοι εξημών. Για την εφαρμογή του κανονισμού υπαριθμό 528 του 2012 σχετικά με τα βιοκτώνα σε ό,τι αφορά τις κατευσουσιοδότηση πράξης. Υπήρξε μια διάταξη του άρθρου 5 που περιλαμβάνει υποχρέωση μέχρι τις 13 Δεκεμβρίου του 2013 να εγκρίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πράξη κατά εξιδιοδότηση που θα ορίζει τα συγκεκριμένα κριτήρια για τις, ε, το ρευματισμό, την κατάργηση χρήσης ενδοκρινικών διαταρακτών. Παρά το γεγονός ότι έχει περάσει πλέον αυτή η προθεσμία, δεν υπάρχει σχετική πράξη καταξιοδότηση από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και επειδή αυτό αποτελεί ένα ζήτημα το οποίο συζητήθηκε ιδιαίτερο εδώ στο Κοινοβούλιο, αλλά και μεταξύ των κρατών μελών και τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι συντονιστέ λοιπόν αποφάσισαν ότι θα έπρεπε να προσκληθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Επιτροπή μα για να εξηγήσει γιατί καθυστέρησε τόσο πολύ αυτή η σημαντική υποχρέωση και να απαντήσει σε οποιοδήποτε τυχόν ερώτημα και καλό θα ήταν, θεωρώ, να δώσουμε το λόγο στον κύριο Μπιόν Χάντσεν, ο οποίος είναι γενικός διευθυντής, ε, μάλλον ε, υπεύθυνο της Επιτροπής, της Αρμόδιας Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκής Επιτροπής, από τη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος. Να μας εξηγήσει λοιπόν γιατί τα σημαντικά αυτά ζητήματα δεν έχουν ακόμα επιληθεί. Έχετε το λόγο. Thank you very much, Mr. Chairman. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη, αξιότιμοι επισκέπτες από τον Bundestag και όλοι οι υπόλοιποι. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας δίνετε αυτή την ευκαιρία να εξηγήσουμε μια ακολουθία γεγονότων που τελικά οδήγησαν ε, την Κομισιόν να λάβει την απόφαση για τη διεξαγωγή μιας εκτίμησης αντικτύπου όσον αφορά την ανάπτυξη επιστημονικών κριτηρίων και την υλοποίησή τους αντί να τηρήσει την προθεσμία που μόλις αναφέρατε που είχε οριστεί στον κανονισμό για τα βιοκτώνα προϊόντα. Το κλειδί των γεγονότων που μας οδήγησε σε αυτή την απόφαση έλαβε χώρα το καλοκαίρι. και μιλάμε για το καλοκαίρι που ήταν καλοκαίρι για όλες τις χώρες από το βορρά μέχρι τον νότο, από τον Ιούνιο μέχρι τον Αύγουστο του 2013. Ήμασταν εντός των χρονών ε, στην ανάπτυξη κάποιων κριτηρίων επιστημονικών για ε, τα επικίνδυνα απόβλητα με σκοπό να εφαρμόσουμε τα κριτήρια αυτά και να αξιολογήσουμε την εφαρμογή τους σε επιμέρους ε, νομοθετήματα. Στους μήνες που προανέφερα συνέβησαν δύο γεγονότα. Πρώτα απ' όλα μια ανακοίνωση προς την Κομισιόν μέσω πολλών οδών ότι οι επιπτώσεις των κριτηρίων που επρόκειτο να εφαρμόσουμε όσον αφορά τη διαθεσιμότητα των χημικών ουσιών στην ευρωπαϊκή αγορά και συνεπώς ε, οι συνέπειες της εφαρμογής τέτοιων κριτηρίων θα ήταν οικονομικά και εμπορικά αρκετά σημαντικές όσον αφορά και το εμπόριο με τους ε, πλησιέστερους εταίρους μας. Πέραν της βιομηχανίας, η οποία μας εξήγησε ότι αυτό που πρόκειται να κάνουμε θα είχε σημαντικές επιπτώσεις, έγινε και μια πολύ σημαντική επιστημονική συζήτηση εκείνους τους μήνες ακριβώς. Τυπώθηκε ένα δημοσίευμα σε πολλές διεθνείς επιστημονικές εφημερίδες και περιοδικά από, τους αρχισυντα... από 18 νομίζω αρχισυντάκτες, αν θυμάμαι καλά τον αριθμό, 18 ή, 18 ή 19 επιστημονικά περιοδικά, όπου αναφερόταν ότι η εργασία της Κομισιόν δεν βασιζόταν σε επιστημονικά στοιχεία και συνεπώς ε, είχε παρουσιάζει κάποιο πρόβλημα. αυτού του είδους την προεδοποίηση λάβαμε από οικονομικούς φορείς και από επιστήμονες και μας οδήγησε σε επαναξιολόγηση της προσέγγισής μας. Χρειάστηκε να επαναξιολογήσουμε την προσέγγιση του κατά πόσο έπρεπε να αναπτύξουμε τέτοια επιστημονικά κριτήρια και μετά να προχωρήσουμε σε συγκεκριμένη αξιολόγηση κάθε νομοθετήματος που αφορούσε την εφαρμογή των κριτηρίων αυτών. Κατά την επαναξιολόγηση αυτή, κατέστη σαφές ε, ότι το 7ο πρόγραμμα για το περιβάλλον που βρισκόταν υπό διαπραγμάτευση μεταξύ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου πρόκειται να καταλήξει σε ένα κείμενο το οποίο είχε συμφωνηθεί μεταξύ των μερών και το κείμενο αυτό περιλάμβανε ως στόχο για το σύνολο της Ένωσης την ανάπτυξη εναρμονισμένων κριτηρίων βασισμένων σε επιστημονικά στοιχεία για τον προσδιορισμό των ενδοκρινικών διαταρακτών και μια σειρά άλλων δράσεων. Εμείς λοιπόν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρήσαμε σκόπιμο λόγω των σημαντικών επιπτώσεων που προβάλλονταν από τη βιομηχανία ως επιχείρημα και από ορισμένους τομείς της βιομηχανίας και λόγω της ε, εκτενούς επιστημονικής συζήτησης που ξεκίνησε εκείνους τους μήνες αλλά και λόγω του σαφούς πολιτικού μηνύματος ε, από το Κοινοβούλιο και από το Συμβούλιο ότι έπρεπε να έχουμε εναρμονισμένα κριτήρια σκεφτήκαμε λοιπόν ότι σκόπιμο ήταν ε, να ακολουθήσουμε μια προσέγγιση αξιολόγηση αντικτύπου για τα εναρμονισμένα κριτήρια και για την υλοποίησή τους σε όλες τις νομοθεσίες ταυτόχρονα. Αυτή λοιπόν ήταν κύριε Πρόεδρε οι τρεις παράγοντες που μας οδήγησαν να περάσουμε από τα συγκεκριμένα κριτήρια και την εφαρμογή της στην ανάπτυξη επιστημονικών κριτήριων και σε εκτίμηση αντικτύπου της εφαρμογής τους σε όλες τις σχετικές νομοθεσίες. Γι' αυτό τον τελευταίο σκοπό αναπτύξαμε έναν οδικό χάρτη, ο οποίος δημοσιεύτηκε περίπου πριν από 6 μήνες ή λίγο περισσότερο. Στον οδικό χάρτη αυτό χαράστε μια στρατηγική και οι επιλογές που επιθυμούμε να αξιολογήσουμε. Ελπίζω αυτό να δίνει τουλάχιστον σε ένα αρχικό στάδιο επαρκείς εξηγήσει ε, για τους λόγους για τους οποίους ε, δεν τηρήσαμε τις ε, καθορισμένες προθεσμίες. Αν έχετε άλλες ερωτήσεις, ευχαριστώ να τις απαντήσω. Ευχαριστώ. Εμείς σας ευχαριστούμε. Και η ώρα των ερωταπαντήσεων. Ο κύριος Στάς έχει ζητήσει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, συνάδελφοι, να ευχαριστήσω τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την απάντησή του. Θα πρέπει να πω ότι πρόκειται για ένα θέμα το οποίο το μας απασχολεί εδώ και πάρα πολύ καιρό. Έχει μεγάλο παρελθόν. Όχι μόνο από το προηγούμενο κοινοβουλίο, αλλά από το προπροηγούμενο, από την προπροηγούμενη σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η ενδοκρινική διαταρακτές έχουν, έχουν πάρα πολύ ε, μεγάλο αντίκτυπο σε χρόνιες ασθένειες, διαβήτη, καρκίνο, προβλήματα αναπαραγωγικά. Και γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν αποφάσισε να αναπτύξει κοινοτική στρατηγική από το 1999 κιόλα. αλλά από τότε δεν έχει μεταφραστεί αυτό σε συγκεκριμένη δράση. Στις διάφορες συζητήσεις τις οποίες κάναμε, για την νομοθεσία για τα βιοκτώνα, όχι στο προηγούμενη θετία, αλλά στην προ-προηγούμενη θετία της έκθεση στην οποία και συμμετείχα γιατί είχα στην αρμοδιότητά μου ένα μικρό κομμάτι της νομοθεσίας εκείνη. Τότε λοιπόν ως κοινοβούλιο αντιταχθήκαμε έντονα στη κριτηρια κάτω. τα οποία ενοχλούν ιδιαίτερως ε, την βιομηχανία και κατά τη διάρκεια της ε, νομοθετικής δραστηριότητας της έκθεσης της ε, κυρίας Μπρέιερ, ως κοινοβούλιο λοιπόν ζητήσαμε πολύ συγκεκριμένα κριτήρια. Σε μια φάση διαπραγμάτευσης με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και με το Συμβούλιο, είχαμε στην αρχή μια φάση 18 μηνών, όπου δώσαμε χρόνο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρουσιάσει πολύ σαφή κριτήρια. Αυτό λοιπόν αρχικά είχε προβλεφθεί για τα τέσσερα χρόνια. Το ίδιο κάναμε και στο προηγούμενη θητεία. Η έκθεση της κυρίας Κλάς, η οποία εγκρίθηκε το 2012, όπου και πάλι ζητήσαμε με σαφήνεια να μας υποβάλει σχετικά κριτήρια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτή λοιπόν η ερώτηση δεν προέρχεται από το πουθενά. Ω Κοινοβούλιο σε διαπραγμάτευση με το Συμβουλίο και σε συζήτηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέσαμε πολύ συγκεκριμένε απαιτήσει, αξιώσει. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αρχικά και το είπε αυτό στην απάντηση ο εκπρόσωπο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε λοιπόν με την κατάρτιση των κριτηρίων αυτών το 2010 αλλά ως Κοινοβούλιο συνεχίσαμε να παρακολουθούμε την διαδικασία όπως και κάνουμε τώρα. Από το 2013 προέκυψε και ψηφίσαμε ένα ψήφισμα για τους ορμονικούς αυτούς διδαράκτες και ζητήσαμε επιστημονικά και οριζόντια ζητήματα προσέγγισης για την ανάπτυξη των κριτηρίων αυτών. Και δηλώναμε πάντα ότι η μελέτη αντικτύπου θα πρέπει να γίνει μόνο εφόσον έχουν οριστεί πρώτα τα επιστημονικά κριτήρια. Αυτή ήταν η γραμμή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τον Ιούνιο του 2013, αγαπητοί συνάδελφοι, μετά από δυόμιση χρόνια εργασία, όλων των αρμόδιων υπηρεσιών, η Γενική Διεύθυνση NV σε μια διαυπηρεσιακή διαβούλευση ξεκίνησε και κατέθεσε μια πρόταση των κριτηρίων και αυτό ήταν πολύ έγκυρα προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία εντό 4 ετών όπω είχε ζητήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τι έγινε λοιπόν τότε. Μπήκε στη μέση η βιομηχανία, Endocrination, μια ταινία. Την έχω εδώ, αν θέλουν να τη δουν οι συνάδελφοι. Εδώ λοιπόν στην ταινία αυτή παρουσιάζεται επακριβώς το τι έγινε. Το Δεκέμβρη λοιπόν το 2013 όταν ξεκινήσε η διαδικασία διαβούλευση, τι έγινε, η εταιρεία Bayer ζήτησε από τον Γενικό Γραμματέα να γίνει διαβούλευση για τα σχετικά κριτήρια. Τι γίνεται μετά. Λίγο αργότερα, στον Ιούνιο, μία ομάδα επιστημόνων αποστέλνει ένα, μία επίστολη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και δηλώνω ότι αυτά που γίνονται δεν συνάδουν με, την επιστημονική, με τα επιστημονικά δεδομένα. 2 Ιουλίου λίγες εβδομάδες αφού το έχει ξεκινήσει η διαδικασία. Και ο χρόνος, ο Κάτριν Ντέις, ο Γενικός Γραμματέας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ξεκινάει άμεσα μια μελέτη αντικτύπου έναν μήνα αργότερα, τον Αύγουστο του 2013. Οι επιστήμονες, οι οποίοι επισταμμένως ασχολούνται με το θέμα αυτό και είναι πολύ ψηλούς κύρους για το θέμα αυτό, δηλώνουν ότι αυτά που έχει γράψει η προηγούμενη ομάδα επιστημόνων, 56 επιστημόνων, δεν είναι ακριβή. Τον Οκτώβριο του 2013, σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, αυτό καταγράφεται και στην ταινία, γίνεται μια συνεδρίαση στο Englobe και τα, οι δύο ομάδες επιστημόνων, οι 56 επιστήμονες, η αρχική και η ομάδα των υψηλά εισταμένων επιστημόνων και αποδεικνύεται ότι η πρώτη ομάδα δεν είχε καθόλου βάση στα σχόλιά της. Ρωτώ λοιπόν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μπορείτε να επιβεβαιώσετε ότι η παρέμβαση από πλευρά της Bayer και η ομάδα των 56 επιστημόνων ήταν καθοριστική σημασία για την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να διεξαγάγει μελέτη αντικτύπου. Δεύτερη ερώτηση. Μπορείτε επίσης να επιβεβαιώσετε ότι οι ενστάσεις των 56 επιστημόνων ήταν πραγματικά χωρίς βάση. Και στη συνεδρίαση που έγινε στην κυρία Γκλόβερ, τα πράγματα διεξήχθησαν, όπως είπα, ένα άλλο στοιχείο στην όλη υπόθεση, η δημόσια διαβούλευση σε ό,τι αφορά τα κριτήρια. Έχουμε το 7ο πρόγραμμα δράσης, έχουμε τον οδικό χάρτη όπου, στον οποίο αναφέρθηκε και ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και είναι πολύ σαφές ότι και τα δύο αυτά έγγραφα δείχνουν προς την κατεύθυνση μιας οριζόντιας προσέγγισης. Οριζόντια προσέγγιση όπου θα εξετάσουμε τις θέσεις αλλά και τα πλεονεκτήματα των ενδεχόμενων δυνατοτήτων. Τον Σεπτέμβριο του 2014 λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε τη διαδικασία διαβούλευση για τα κριτήρια αυτά για του ε, διαταράκτες και τι διαπιστώνουμε ότι δεν πρόκειται για οριζόντια προσέγγιση. Περιοριζόμαστε στα βιοκτώνα και στα ζυζανιοκτώνα, ενώ ξέρουμε ότι πολλά περισσότερα περιλαμβάνονται. Θα πρέπει να κοιτάξουμε και την νομοθεσία για το είδωρ, για τα καλλιντικά και η διαβούλευση περιορίζεται στον οικονομικό-κοινωνικό αντίκτυπο και όχι σε ενδεχόμενα α, ωφέλη πλέον εκτίματα των διαφόρων κριτηρίων. Και νομίζω λοιπόν αυτά που συμβαίνουν αυτή τη στιγμή είναι αντίθετα με το έβδομο πρόγραμμα δράση και με την οδικό χάρτη. Πώ θα φροντίσετε λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υπάρχει οριζόντια προσέγγιση σε ό,τι αφορά τα κριτήρια αυτά και να λεφθούν υπόψη και τα πλέον εκτίματα των διαφόρων δυνατοτήτων. Και τέλος, πότε ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή σκοπεύετε να υποβάλλετε πράξεις κατά εξουσιοδότηση για το θέμα αυτό, γιατί θεωρώ ότι ο χρόνος πιέζει. E Ευχαριστούμε. Δίνουμε το λόγο στον συνάδελφο, τον κύριο Γκρότε. Σας ευχαριστώ. Ο Μπάρτ Στάσε πάρα πολλά είπε που ήθελα να πω κι εγώ. Το όλο θέμα μας απασχολεί από το 2008 σε ό,τι αφορά τις διαπραγματεύσεις για τα διδανειοκτώνα, όπου διευκρινίσαμε σε ό,τι αφορά τα κριτήρια ότι θέλουμε κάτι συγκεκριμένο. Το 2013 ήταν λοιπόν, τέλη 2013 έλεγε η προθεσμία. Πέντε χρόνια καιρό είχανε. Και για τα εκτώνα είχαμε κάνει σχετική αίτηση. Για μας είναι σαφές. Υπάρχει εντύπωση ότι όλα αυτά αναβλήθηκαν μετά από πίεση ενός πολύ ισχυρού λόμπι. Αυτή είναι η εντύπωση που δημιουργείται και ίσως θα μπορούσατε να μας τα παρουσιάσετε όλα αυτά ίσως υπό κάποιο άλλο πρίσμα. Αλλά αυτή είναι η εντύπωση που μας δείτε. Το θέμα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για το Κοινοβούλιο και με διάφορες ε, οδηγίες νομοθετήσαμε και από πλευρά Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχουμε τίποτα ακόμα συγκεκριμένο στα χέρια μα. Είμαστε και περιμένουμε ακόμα. Κατά πόσο θα το ανεχτούμε αυτό, πραγματικά πρέπει να το διαβολευτούμε ή κατά πόσο θα πρέπει να κινητοποιηθεί και το Κοινοβούλιο για να υποστηρίξει κάποια ζητήματα τα οποία δεν έχουν ολοκληρωθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αλλά ίσως να μπορέσετε να μας δώσετε κάποια εξήγηση. Εγώ πραγματικά ε, είμαι έκπληκτος που χρειάστηκε τόσο πολύ χρόνος, παρά το γεγονό ότι είναι στην κορυφή των προτεραιότητων του Κοινοβουλίου το θέμα αυτό. Ευχαριστούμε πολύ. Ο συνάδελφος κ. Πενδύ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν θα επαναλάβω αυτά τα οποία είπαν οι τη συνάδελφοι Τάση και Χρόντα, αλλά έχω μια ερώτηση να υποβάλω, αλλά και μια παρατήρηση. Παρατήρηση πρώτα. Όλοι γνωρίζουμε ότι οι προτάσεις είχαν ετοιμαστεί από την ε, αρμόδια Διεύθυνση της Επιτροπής και πρόκειται περί πολιτικής αποφάσεως που απέτρεψε την δημοσιοποίηση των προτάσεων αυτών. Και αφού πρόκειται για πολιτική απόφαση και ο υποψήφιος πρόεδρος ο κ. Γιούνκερ αποφάσισε ότι το σώμα των επιτρόπων είναι πολιτικό όργανο και είναι η Επιτροπή Πολιτική. Μου φαίνεται πάρα πολύ παράδοξο το ότι εδώ συζητούμε με υπαλλήλου τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή γιατί Το μέλλον νομίζω ότι θα πρέπει η συζήτηση να γίνεται με μέλλον, μέλο συγγνώμη τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή με έναν επίτροπο που αυτό είναι ο πολιτικά υπεύθυνο. Οπότε η πολιτική απόφαση αυτή που ήταν τροχοπέδη σε όλη τη διαδικασία να συζητηθεί. Οπότε θα πρέπει μια που είναι απλά και ο Γενικό Γραμματέα να τα συζητήσουμε με τον ε, πρόεδρο Μπαράσο και στο μέλλον τον κύριο Γιούγκερ. Έτσι νομίζω πρέπει να δουλεύουμε εδώ εφόσον είναι πολιτική. Και ε, τότε θα πρέπει να συζητούμε ως πολιτικοί εμείς με εκείνους. Έχω να ρωτήσω το εξής. Όλα αυτά αφορούν επιστημονικά κριτήρια. Μας είπε ο υπάλληλος Επιτροπής ότι οι επιστήμονες αμφισβητούν την επιστημονική τεκμηρίωση των προτάσεων και αν έχει δίκιο στην άλυση του ο κύριος Στάς, τότε αυτά τα επιχειρήματα ήταν έολα. Οπότε, αφού ζητούμε επιτυμονικά κριτήρια και οικονομικές επιπτώσεις, ε, τότε τη στιγμή αυτή αυτά δεν έχουν σημασία. Και αν συζητούμε λοιπόν για το background το επιστημονικό, άρα θα πρέπει να δούμε σε αυτή την πορεία της εξέτασης των επιστημονικών τεκμηρίων ε, γιατί να πρέπει να ζητούμε την επιστημονική αξιολόγηση γιατί αυτό να μην γίνει εκ των υστέρων γιατί υποτίθεται ότι η επιστημονική τεκμηρίωση είναι ξεκάθαρη και επομένως αυτό το οποίο θα έχει μετά σημασία θα είναι οι επιπτώσεις οι οικονομικές. Άρα μήπως μπορεί αυτό να μας απαντήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ πολύ. Το λόγο έχει συνάδελφος κ. Yeah. Uh, uh, Ευχαριστώ πολύ. Συμφωνώ με τα όσα υπόθηκαν. Χρειαζόμαστε μια καθαρή πολιτική συζήτηση. Γιατί αν λαμβάνονται τέτοιε αποφάσει κατά των όσων αποφασίσαμε εμεί εδώ και κατά του 7ου περιβαλλοντικού προγράμματο, παραβλέποντα τα όσα κάναμε εδώ, και παραβλέποντας και επιστημονικά στοιχεία, πέρυσι στη Δανία, στις αρχές του, του έτους, κανείς δεν έχει αμφισβητήσει τα επιστημονικά στοιχεία ότι οι επιπτώσεις είναι πολύ σοβαρές για τα γέννητα βρέφη και Επίσης ότι οι επιπτώσεις ε, στην ανδρική γονιμότητα είναι πολύ σημαντικές και αποδεδειγμένες. Πρέπει να κάνουμε λοιπόν κάτι. Απλά θα ήθελα να προσθέσω επίσης ότι πρέπει να υποστηρίξουμε τη Σουηδία η οποία ζήτησε ε, ε, κατέγγειλε στο δικαστήριο την Κομισιόν για την παραβίαση της νομοθεσίας και για μη τήρηση των υποσχόμενων. Είναι εξωφρενικό ότι η βιομηχανία μπορεί να ασκήσει τέτοιες ποιώσει μέσω των λόμπι της και να λέει ότι δεν θα εξυγχρονίσει την παραγωγή της και ότι θα συνεχίσει χωρίς να ενδιαφέρεται καθόλου για το ποιες είναι οι επιπτώσεις για τα αγέντα βρέφη μας και για όλους τους υπόλοιπους. Πρέπει να κάνουμε κάτι εδώ. Πρέπει να υποστηρίξει αυτή η Επιτροπή τη Σουηδία και να κάνει κάτι. Και να σταματήσουν να μας μπλοκάρουν ξανά και ξανά. Ευχαριστούμε. Δεν βλέπω να ζητάει κάποιο άλλο το λόγο από του συναδέλφου. Να δώσω λοιπόν το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να απαντήσει. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. Στα γερμανικά, στα ολλανδικά και στα δανέζικα Ευχαριστεί πολύ ο κύριος ομιλητής ε, για τις ερωτήσεις και θα κάνω ό,τι μπορώ για να αναλύσω και να εξετάσουμε περισσότερο και να απαντήσω, ελπίζω, ικανοποιητικά στις ερωτήσεις. Το ευκολότερο για να ξεκινήσω είναι τα δύο αποφασιστικά ζητήματα μπορώ να σας επιβεβαιώσω με βεβαιότητα ότι το πλήθος των μηνυμάτων που λάβαμε από τη βιομηχανία και που οδήγησαν στα γεγονότα του καλοκαιριού του 2013 ήταν ένας από τους αποφασιστικούς καθοριστικούς παράγοντες που οδήγησαν την Κομισιόν να πραγματοποιήσει ε, ε, εκτίμηση αντικτύπου των ε, επιστημονικών κριτηρίων και της εφαρμογής τους σε πολλά και διαφορετικά νομοθετήματα. Να τονίσω ότι το ένα email ε, στο οποίο αναφερθήκαμε ήταν απλά ένα από τα μηνύματα που έλαβε η Κομισιόν αλλά σίγουρα συνέβαλε στο να αποφασίσουμε εμείς στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι ήταν απολύτως αναγκαίο να εξετάσουμε το την αξιοπιστία των ισχυρισμών της βιομηχανίας. Μετά υπήρξε και άλλο ένα καθοριστικό ζήτημα, το ζήτημα των 56 ε, επιστημόνων ή συντακτών αρκετά μεγάλου αριθμού διεθνών επιστημονικών περιοδικών. Και ναι, μπορώ να σε βεβαιώσω ότι χάρη στη συνάντηση με τον Επιστημονικό Σύμβουλο του Πρόεδρου καταφέραμε να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι τα ζητήματα που έθιξαν αυτοί οι διακεκριμένοι επιστήμονες είναι ζητήματα που είναι γνωστό ότι είναι αβέβαια επιστημονικά και ότι δεν είναι τόσο σημαντικά για τα ίδια τα κριτήρια. Πρέπει να σας πω ότι αυτοί οι διακεκριμένοι επιστήμονες των ε, διεθνών επιστημονικών περιοδικών στα άρθρα τους ε, ξέχασαν ή παρέβλεψαν μια αναφορά στο έργο της Κομισιόν που θεωρούσαν ότι είναι μη επιστημονικό. Οπότε η παρεβλεψαν μια αναφορα στο εργο το εισκομισιων που θεωρουσαν οτι ειναι μη επιστημονικο οποτε η Κομισιόν δυσκολεύτηκε να καταλάβει τι δυσαρεστούσε αυτούς τους επιστήμονες ε, όσο το κύριο Σεγκλόβρο επιστημονικό Σύμβουλος κάλεσε, συνάντησε. Αλλά το γεγονός και μόνο ότι τόσοι πολλοί συντάκτες ε, διεθνών επιστημονικών ε, περιοδικών έγραψαν τόσο αυστηρά άρθρα επικρίνοντας τόσο αυστηρά το επιστημονικό έργο της Κομισιόν το οποίο προσπέγραφαν επίσης και πολλοί άλλοι διεθνείς επιστήμονες, οδήγησε την Κομισιόν στο να αποφασίσει ότι ήταν αναγκαίο να αξιολογηθούν τα αιτήματα αυτά και το πόσο ήταν ευλόγα. Χάρη στο έργο της κυρίας Αγγλόβερ ε, και χάρη στη συνεδρίαση που κάλεσε με όλους αυτούς τους επιστήμονες μέσα σε μια μέρα η οποία κατέληξε σε πολύ σαφή συμπεράσματα σήμερα λοιπόν χάρη σε αυτή τη συνάντηση μπορούμε να πούμε σήμερα ότι τα ζητήματα επιστημονικής αβεβαιότητας που συμφωνήθηκαν σε εκείνη τη συνάντηση είναι ζητήματα τα οποία γνωρίζουμε εδώ και κάποιο καιρό και εγώ ε, εργάζομαι εδώ από τότε που υιοθετήθηκε η στρατηγική του 1999 και προσπαθούμε να τα διασαφηνίσουμε. Τώρα αν δούμε την εκτίμηση αντικτύπου και τον οδικό χάρτη και την πρόσφατα δημοσιευθήσα ε, δημόσια διαβούλευση θα δείτε στον οδικό χάρτη ότι η πρόθεσή μας είναι να αξιολογήσουμε τα πλέον εκτήματα και τα κόστη. Πρόθεσή μας είναι να αξιολογήσουμε τις επιπτώσεις οριζόντιων κριτηρίων σε όλες τις νομοθεσίες και ειδικότερα στα έξι νομοθετήματα τα οποία αναφέρουν ρητά τους ενδοκρινικούς διαταράκτες. Και αυτή είναι η πρόθεσή μας. Όσον αφορά τις ερωτήσεις ε, της δημόσιας διαβούλευσης, έγιναν αρκετέ συζητήσεις για το κατά πόσο η διαβούλευση έπρεπε να είναι πολύ ευρεία με πολλές ερωτήσεις ή στοχευμένη στους τομείς κλειδιά για τους οποίους θέλαμε πληροφορίες. Και τελικά θεωρήσαμε ότι η δεύτερη λύση ήταν πιο ωφελημή για μας ε, και για ε, να μην σπαταλά το χρόνο των όσων απαντήσουν τις ερωτήσεις. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρόκειται να δούμε την ίδια την, ε, στην εκτίμηση αντικτύπου τα ωφέλη. Μάλιστα σκοπεύουμε να αναθέσουμε μέσω σύμβαση ε, ε, την αξιολόγηση των πλέον εκτιμάτων. Και φυσικά αυτό δεν σημαίνει ότι θα ξεχάσουμε την αξιολόγηση του οριζόντου χαρακτήρα των κριτηρίων. Στη συνέχεια έλαβα την ανοιχτή ερώτηση, την ανοιχτή ερώτηση που θα μου περιορίσει να παρουσιάσω κάποια σχετική εικόνα των πραγμάτων. Έχουμε δύο ροές ισχυρισμών ε, για σημαντικές επιπτώσεις και για σημαντικές ε, επιστημονικές αβεβαιότητες. Εμείς ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ως Δημοσιολειτουργή, θεωρήσαμε υποχρέωση μας να διερευνήσουμε το κατά πόσο είναι αξιόπιστοι οι ισχυρισμοί αυτοί. Οι επιστημονικοί ισχυρισμοί, όπως είπα, στο μεταξύ έχουν επιληθεί το ζήτημα της σημαντικής επίπτωσης ε, στη βιομηχανία είναι κάτι που πρόκειται να διαπιστωθεί και να εξεταστεί με την εκτίμηση αντικτύπου που αυτή τη στιγμή δεν εργούμε. Τώρα, γιατί κάνουμε εκτίμηση αντικτύπου επιστημονικών κριτηρίων. Να ξαναναφερθώ στον οδικό χάρτη. Στον οδικό χάρτη μπορείτε να δείτε ότι έχουμε πολλές επιλογές οι οποίες σχετίζονται με τα επιστημονικά κριτήρια. Οι δύο εναλλακτικέ που σχετίζονται με τα επιστημονικά κριτήρια είναι αν θα συμπεριλάβουμε ή όχι κατηγορίε. Αυτό ήταν κομμάτι τη έκθεση ίδια πρωτοβουλία του Κοινοβουλίου πέρυσι ότι όντω θέλατε κατηγορίε, αλλά εμεί πρέπει να δούμε στην εκτίμηση αντικτύπου μα αν πρέπει να συμπεριληφθούν ή όχι κατηγορίε στα επιστημονικά κριτήρια. Και μετά υπήρχε το άλλο στοιχείο, και εδώ τα πράγματα είναι λίγο πιο τεχνικά, το ζήτημα Ε, σχέσεις του potency, του, της σημαντικότητας και εμείς πρέπει να δούμε κατά πόσο αυτό το στοιχείο πρέπει να συμπεριληφθεί ή όχι στα κριτήρια ως κομμάτι των επιλογών πολιτικής. Όπως βλέπετε λοιπόν υπάρχουν εναλλακτικές σε σχέση με τα επιστημονικά κριτήρια Υπάρχουν επιλογές ε, και για τα ωφέλη και τα πλεονεκτήματα και το πλήρες πακέτο αυτό θέλουμε να αξιολογήσουμε. Δεν θα σχολιάσω άλλο εκτός αν υπάρχουν και άλλες ερωτήσεις. Ευχαριστώ. Ε, Ευχαριστούμε. Μπορούμε να περάσουμε λοιπόν στο επόμενο σημείο πριν περάσουμε στο επόμενο σημείο να σα ε, χαιρετήσω τις εκπροσώπους ε, της Επιτροπής Γενικών Τρεβίζο που έχουν έρθει εδώ πέρα. Το επόμενο σημείο έχουμε αλλάξει τα σημεία της ημερήσιας διάταξης οπότε τώρα μιλάμε για τη δυνατότητα που έχουν τα κράτη-μέλη να περιορίζουν ή να απαγορεύουν την καλλιεργία γενικτικών τροποποιημένων οργανισμών στην επικράτειά τους. Όπως ε, γνωρίζουμε όλοι, αυτή η πρόταση βρίσκεται υπό εξέταση εδώ και πάρα πολύ καιρό. Η Κομισιόν έκανε την πρότασή της τον Ιούλιο του 2010 και το Κοινοβούλιο τον Ιούλιο του 2011 υιοθέτησε σε πρώτη ανάγνωση τη θέση του. Το Συμβούλιο 12 Ιουνίου του 2014 κατέληξε σε πολιτική συμφωνία η οποία μας κοινοποιήθηκε στην πρώτη σύνοδο μετά το καλοκαίρι στο Στρασβούργο. Έτσι λοιπόν μπορούμε να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας για διαπραγματευτική εντολή. Δίνω αμέσως το λόγο στην εισηγήτρια, την κυρία Φρέντερη Κρίς για την ομιλία της. Παρακαλώ. Merci, Monsieur le Je suis je γιατί αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να έχω 6-7 λεπτά. Να είμαι σύντομη, αλλά αφού είχε τόσο πολύ το ζήτημα, ε, νομίζω ότι θα πρέπει να μπορέσουμε μετά από τόσους χρόνια δουλειάς να δούμε τι θα γίνει και τι θα γίνει και με τον τριμερή διάλογο. Οπότε είπαμε ότι πρόκειται τώρα για ένα κοινό σημείο το οποίο το τόνισαν όλοι στην πρώτη ανταλλαγή χωρίς να είχαμε έγραφο τότε αρχές Σεπτεμβρίου. Και πρόκειται για τη διαχείριση σε ευρωπαϊκό επίπεδο για το τι γίνεται με τους γενικά τροπημένους οργανισμούς. Να πρέπει να δούμε ποιος είναι ο πιο φυσικός τρόπος ε, γιατί θα πρέπει είπαμε να γίνει η, κάποιο είδους ανάθεση, εκχώρηση δικαιωμάτων και άρα θα πρέπει να δούμε αν μπορούν τα κράτη-μέλη να περιορίζουν ακριβώς την καλλιέργεια των ε, ε, οργανισμών αυτών στην επικρατεία τους. Τον Ιούλιο, ε, επίσημο και επιτροπή, είχαμε κατόπιν και τις ακροάσεις, όπου συμμετέχουν όλες οι πολιτικές ομάδες και όλοι είπαν θα πρέπει να γίνει μια μεταρρυθμίση σε βάθος και να δούμε τι θα γίνει με την διαδικασία λήψη αποφάσεων για την ε, αδειοδότηση, για την καλλιέργεια των οργανισμών αυτών. Και ο Ζήλ αξιολογεί με το θέμα και κατέληξε στα ίδια θέματα μαζί, ο συνάδελφος Ζήλ. Και είπαμε και οι δύο ότι χρειάζεται περισσότερη ευελιξία. Να έχουν τα κράτη-μέλη περισσότερη ευελιξία, ε, ώστε να μπορούν να εξασφαλίσουν την ασφάλεια δικαίου. Και γι' αυτό και έχουμε την τροποποίηση της οδηγίας του 2001 για τους οργανισμούς αυτούς, κάτι το οποίο έχει επανειλημμένα ε, συζητηθεί. Ε, ε, αυτό το θέλει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και συμφωνεί η μεγάλη πλειοψηφία των Ευρωβουλευτών. Ξεκινήσαμε τον Ιούλιο 2001 για αυτή την πορεία και πλειοψηφία ήταν συντριπτική, υπήρχαμε τότε υπέρ αυτής πρότασης 548 ψήφους, οπότε και εγώ έλαβα αυτή την ε, εντολή, αλλά το ήθελε και το Συμβούλιο να προχωρήσουμε, όταν ε, τοποθετήθηκε στις ε, ε, αρχάς του θέρους για αυτή την πρόταση του Ιουλίου. Έχουμε εδώ τώρα κάποιες τροπολογίες, αλλά θα πρέπει να σας πω ότι η θέση του Συμβουλίου νομίζω ότι θα πρέπει να βελτιωθεί για να δούμε επομένω τι γίνεται για αυτή την περίφημη πρώτη φάση ε, όσον αφορά την ε, θέσπιση αυτής της νέας ε, διαδικασία τη αυτοεξέρευσης. Για, είπαμε εδώ πέρα είναι η θέση του Συμβουλίου για τη φάση αυτή της αδειοδότησης, για την άδεια καλλιέργειας αυτών των ε, τρόπινων οργανισμών και είπαμε ότι υποχρεωτικά θα πρέπει να περάσουμε από αυτή την πρώτη φάση και μέσω της Επιτροπής θα πρέπει να υπάρξει αυτή η αίτηση από κάποια επιχείρηση και η χώρα αυτή δέχεται την αίτηση για την αδειοδότηση και κατόπιν τα κράτη-μέλη ενεργοποιούν τη δεύτερη φάση όσον αφορά το αν θα επιτραπεί ή όχι σε εθνικό επίπεδο και με κάποια ε, ε, κριτήρια οικονομικά, γεωργικά κλπ. λαμβάνει η απόφαση. Κατά αυτή τη δεύτερη φάση που είναι του κυρίως φάση για την συζήτηση. Επομένως με ενδιαφέρει πολύ το Κοινοβούλιο και εγώ και άλλοι έχουμε ε, κάποιες επιφυλάξεις για την αποτελεσματικότητα αυτών των νέων μηχανικών. Ε, μας έδωσε ευγενώ η Κομισιόν κάποιες εξηγήσει, αλλά δεν ήρθησαν οι απορίες μας. Ακόμα βέβαια μιλούμε για βιοκτώνα αλλά όσον αφορά τους γενετικά τρομερούς οργανισμούς δεν έχει ακόμα δοκιμαστεί αυτή η καινούργια διαδικασία σε αυτό το καυτό θέμα. Χρειάζεται επομένω κάτι το που να είναι στεγανό νομικά και θα πρέπει και τα κάτι μέλη να μπορέσουν να δικαιολογήσουν τι γίνεται. Και εδώ παραδείγματος τροπολογία 22. Επομένως, αιτιολόγηση επί βάση των προαναφερθέντων κριτηρίων για την ασφαλεία του δικαίου, αλλά επίσης για να έχουμε και διαφάνεια σε επιδοκρατών μελών, θα πρέπει τα κρατημέλη να μπορούν να παρατείνουν το σχετικό διάστημα, σχετική προθεσμία. Εδώ προβλέπονται στο κείμενο 30 ημέρες. Ε, Βεβαίω, δεν έχω καταλήξει, διάβασε την επικοινωνία ο οποίος μας είπε από πλευρά ε, συμβουλίου τη δική του εμπειρία, ε, με κάποια επιχειρήματα, οπότε και είμαστε έτοιμοι να τον ακούσουμε. Πάντως, όσον αφορά στη δεύτερη φάση, τον υπουργικό χαρακτήρα και την ενεργοποίηση διαδικασίας, αφού περάσει κανείς από την πρώτη φάση. Επομένως, de facto τώρα, η δεύτερη φάση όμως λαμβάνει περιφερειακό χαρακτήρα, ενώ είναι πάρα πολύ σημαντική για, για το έργο μας. Κατά αυτό αντιβαίνει με τους βασικούς σκοπούς της οδηγίας, δηλαδή να υπάρχει περισσότερη ευελιξία ενέργειας ουράς κρατών μελών. Ε, σας παραμένω τώρα στην τροπολογία 24, που ε, από την αρχή αρχή λέει ότι αυτά όλα δεν, δεν ε, κριτήρια και σαν δεύτερη επιλογή τα κράτη-μέλη και επομένως σας παραπέμπω σε αυτές τις προτάσεις επί τη βάση της πρότασης του 2012 επί Δανέζικης Προεδρίας. Και με την ευκαιρία έχω μια ερώτηση για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή επανειλημμένα. Μας λέτε ότι θέλετε να διευρύνετε τα εργαλεία που έχουν στα χέρια τους τα κράτη-μέλη. Δεν νομίζετε ότι με αυτή την προσέγγιση, σύμφωνα με την τροπολογία 24, ε, καλύπτω καλύτερα την αρχική σας πρόταση του 2010 σε σχέση και με την τωρινή θέση του Συμβουλίου. Τρίτον, κάτι το οποίο αφορά ε, την φάση 2 και όχι την ε, σχέση των δύο φάσεων. Διαβάζουμε το κείμενο του Συμβουλίου και βλέπουμε ότι το πιο βασικό για μας ε, γίνεται τώρα συμπληρωματικό περιθωριακή σημασία. Επομένω, εντό δύο ετών μετά την ημερομηνία χορήγηση κλπ. κλπ. Λέει. Και έχουμε αυτή την καινούργια διαδικασία του άρθρου 5 και λέει εδώ το κρατό μέλος θα πρέπει να ξέρει ακριβώς ε, πώς, είναι οριοθετημένη η καλλιέργεια των ε, γενετικά τρομένων οργανισμών. Μην ξεχνάμε ότι εδώ ο σκοπός είναι η ασφάλεια δικαίου. Σα παραμπέμπω στις τροπολογίες 25 και 26, όπου ο σκοπός είναι να έχουμε μια διαδικασία πιο ασφαλή, πιο στεγανή και πιο συνεπή. Είναι ξεκάθαρη η εντολή που μου έχει δώσει το Κοινοβούλιο στην προηγούμενη θητεία. Γιατί οι περισσότερε τροπολογίε στι οποίε σα παραπέμπω αφορούν κάποια σημαντικά σημεία που συγκέντρωσαν τη συνένεση τη μεγάλη πλειοψηφία των βουλευτών. Και τώρα έχουμε την περίφημη λίστα των ε, grounds, στην αγγλικά, των κριτηρίων, των, των ε, που αφορά την τροπολογία 25 και έχουμε τη δουλειά της Κορίν ε, Λεπάς του 2011. Και εδώ έχουμε ακριβώς αυτή τον συμπληρωματικό χαρακτήρα των κριτηρίων που μπορεί να επικαλεστεί το κράτος μέλος. Και έτσι δικαιολογείται η αλλαγή της νομικής βάσης. Και εδώ σας παραδείγμα στην τροπολογία μου, σύμφωνα με την πρώτη ανάγνωση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εδώ έχω προσθέσει ένα καινούριο στοιχείο σημαντικό ότι το κράτος μέλος επί τη βάση της διαχείρισης του κινδύνου θα πρέπει από τη μία να απευθύνεται στην ΕΦΣΑ και από την μεριά στο, η Κομισιόν πρέπει να απευθύνεται στο κράτος μέλος που διαχειρίζεται λοιπόν τον κίνδυνο. Και για να έχουμε τώρα περισσότερη ασφάλεια και πιο δίκαιη ρύθμιση να σας πω με δύο λόγια τι γίνεται με τις υπόλοιπες τροπολογίες. Ήδη το Σεπτέμβριο είπαμε για την συνύπαρξη για, τα, για μη γενικατροπημένους και γενικατροπημένους οργανισμούς. Τα έχουμε πει λοιπόν στην ανταλλαγή απόψεων. Μετά στο τροπολογία 29, είναι πολύ σημαντικό, ο Ριπένον πληρώνει, αυτή η γνωστή αρχή, τα κριτήρια προβλεψιμότητος, ε, σημαντικά επίσης και στο αυτό στις τροπολογίες μετά 30 και 31 που στο κείμενο ε, μνημονεύω τον κανόνα της διαφάνειας ακριβώς όπως προβλέπετε. Και ε, μακρηγόρησα, αλλά τέλος πάντων τώρα τη σκητάλη συνάδελφοι. Το σημαντικότερο για μας τώρα είναι ότι ξέρουμε σε ποια σημεία διαφωνούμε και σε ποια συμφωνούμε. Αλλά σημαντικό είναι στην πρώτη συνάντηση του τριμερούς διαλόγου να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε μια τοποθέτηση ε, οι εισηγήτρες και όλοι οι συγχυτές και στον χρόνο που προβλέπετε, στον χρόνο που να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε το έργο μας. Κώστιντες. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστούμε και την κυρία Ρης ε, για τις προτάσεις και συστάσεις της. Στην τελευταία συνεδρίαση εδώ στην Επιτροπή αντιληφθήκαμε ότι το ζήτημα αυτό είναι επίγον. Και ζήτημα για το οποίο ο καθένας έχει κάποια διαφορετική γνώμη. Καλωσορίζω τις προτάσεις της εισηγήτριας και ειδικότερα το γεγονός ότι η κυρία Ρης προτείνει στα κράτη-μέλη τα κράτη-μέλη να μπορούν να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα για την αποφυγή μη επιθυμητών ή τροποποιημένων οργανισμών σε συγκεκριμένες περιοχές και να περιορίζουν τη διαδοσή τους. Είναι σημαντικό σημείο αυτό του κειμένου. Τώρα κάτι ενημερωτικό. Συμφωνώ απόλυτα με την εισηγήτρια. Το ίδιο ισχύει και για την εκτίμηση δικτύπου εδώ για την πρόταση του 2010. Οι δοκιμές αυτές είναι δεσμευτικές. Και πιστεύω ότι θα έπρεπε να είμαστε σκληροί και ακαμπτοί όσον αφορά αυτό το σημείο. Έχω λίγο διαφορετική άποψη όσον αφορά την αξιολόγηση κινδύνου. Όσον αφορά τη γενική αξιολόγηση κινδύνου για το περιβάλλον και την υγεία, δεν συμφωνώ απόλυτα με τη διατύπωση εδώ. Να σας υπενθυμίσω ότι εδώ συζητάμε μια οδηγία η οποία δίνει στα κράτη-μέλη την ελευθερία να αποφασίζουν ε, για μερική ιονική απαγόρευση. Εγώ δεν θεωρώ ότι αυτό είναι το σωστό μέσο το να αρχίσουμε να αλλάζουμε τις ε, διαδικασίες εξολόγησης κινδύνου. Θα έπρεπε αυτό να εντάσσεται αντίθετα στην ε, διαδικασία εξουσιοδότησης. του Ζαν Κλοντ Γιούνκερ πρότεινε αναθεώρηση αυτού αλλά δεν είναι αυτός ο σωστός τρόπος ε, για να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα αυτό. Με τη διαδικασία την ε, δύο επιπέδων, γιατί αυτό ε, αποτελεί και την ουσία της πρότασης της κυρίας αλήφθησε η απόφαση βάσει της πρότασης του Συμβουλίου του 2012. Εγώ συμφωνώ σε οτιδήποτε δίνει πιο πολλέ αρμοδιότητε στα κράτη-μέλη για να μην εφαρμόζουν τη γενετικώ ε, τροποποιημένα προϊόντα, αλλά τι, πρόκειται, τι προτίθεται να κάνει η κυρία Ρης για να πετύχουμε να περάσει αυτή η πρόταση μετά το 2012 σε ό,τι αφορά τον κατάλογο των ε, αιτιολογιών. Εδώ βρίσκουμε τα πράγματα αρκετά θετικά, ιδιαίτερα τις προτάσεις για το κοινωνικό αντίκτυπο και σε ό,τι αφορά τον ε, αγροτικό αντίκτυπο. Είναι βελτιωμένη οι προτάσεις, αλλά θεωρούμε ότι δεν υπάρχει επαρκής ε, ε, και επακριβής διευκρινήση και ότι εξακολουθούν να περιορίζονται πολύ τα δικαιώματα των κρατών μελών. Θα πρέπει να υπάρχουν επαρκείς αιτιολογίες για να αρνούνται τα κρατημέλη τα γάμματα ομικρών σε ό,τι αφορά τώρα το άρθρο για ε, την ε, τεχνολογία των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών. Μας εξήγησαν γιατί οι κανόνες για την ενιαία αγορά χρησιμοποιήθηκαν και γιατί η νομική βάση τροποποιήθηκε στο σημείο αυτό. Θα ήθελα λοιπόν να μας πει η εισηγήτρια γιατί αναφέρει τον τομέα του περιβάλλοντος και Τέλος, μία παρατηρήση. Οι συστάσεις αυτές είναι απαραίτητες για να υπάρχει επιτέλους και κάποια νομική βεβαιότητα σε ό,τι αφορά την καλλιέργεια γαμματάλφα ομικρών. Και προκειμένου να μην υπάρχει αυτή η αβεβαιότητα στα κράτη-μέλη. Η αβεβαιότητα που είναι ένα έντονο στοιχείο σήμερα. Ευχαριστούμε ο Αντιπρόεδρος κ. Σπαρνιό. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, πρώτα απ' όλα θα ήθελα να χαιρετήσω το έργο της εισηγητριάς μας, της κυρίας Φρεντερικ Ρίς. Μας παρουσίασε σήμερα μια πολύ ολοκληρωμένη και ισορροπημένη έκθεση που εκφράζει την θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε πρώτη ανάγνωση. Πρέπει να το υπενθυμίσουμε αυτό. Σε αυτή την έκθεση βρίσκουμε τις περισσότερες προτεραιότητες που έχουμε προασπίσει η ομάδα των σοσιαλιστών και δημοκρατών ε, τις αιτίες απαγόρευσης, ε, την αναγκαιότητα δεσμευτικών μέτρων συνύπαρξης ώστε να αποφευθούν οι μολύνσεις των παραδοσιακών καλλιεργιών από γενετικώς τροπημένες καλλιέργειες, η ενίσχυση της μεθόδου αξιολόγησης των κινδύνων από την ΕΦΣΑ και μεγαλύτερη διαφάνεια στη διαδικασία απαγόρευσης. Ε, από τις νέες τροπολογίες προτείνει η κυρία Ρής, ε, υποστηρίζω αυτές που επιτρέπουν στα κράτη-μέλη να τεθούν σε καλλιέργεια για τα 10 χρόνια που διαρκεί η ευρωπαϊκή εξουσιοδότηση των πηγαμών μικρών. Αναφέρομαι στις τροπολογίες 17, 19, 25 και 26 που παρέχουν μεγαλύτερη ευελιξία στα κράτη-μέλη και ενισχύουν την ασφαλεία δικαίου της πρότασης. Επίσης βλέπουμε πολύ ευνοϊκά τις τροπολογίες 10 και 22 που εισάγουν την αναγκαιότητα ε, για ένα κρατό μέλο να αιτιολογήσει απόλυτα το αίτημα το απαγόρευση καλλιέργειας ενός γενετικού στροπημένου οργανισμού από τη φάση 1 και όχι πλέον στη φάση 2. Θα ήθελα να κάνω όμως μια ερώτηση στην εισηγητριά μας, τη Φρεντερικ Κρίς. Τα κράτη-μέλη θα μπορούν να αιτιολογήσουν ε, το αίτημα απαγόρευσης τους στη φάση 1 ενώ δεν θα έχουν ήδη λάβει όλες τις πληροφορίες από τον Ετούντα την επιχείρηση των γενετικοστροπημένων οργανισμών. Επίσης, ε, για να ενισχύσω τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα υποβάλω τροπολογίες για τα ακόλουθα θέματα. Πρώτη τροπολογία για την επισήμανση χωρίς πήγαμα όμικρον ώστε να αποφευθούν διαστρεβλώσεις του ανταγωνισμού, οι γεωργοί θα πρέπει να μπορούν να ανατρέξουν σε επισημάνσεις απουσίας γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών στα προϊόντα τους. Δεύτερη τροπολογία αφορά τις προσθήκες στον κατάλογο αιτιών περιορισμού ή απαγόρευσης. Διατήρηση της λίστας αιτιών δημόσιας τάξης και την αναγκαιότητα αποφυγής ύπαρξης των γενικών τροποποιημένων οργανισμών σε άλλα προϊόντα καθώς ε, θα, ε, επίσης θα προσθέσω και ε, αιτίες που αφορούν την κοινή γνώμη βάσει των αποτελεσμάτων δημοψηφισμάτων. Τέλος, η τεχνολογική έρευνα ώστε να δούμε τους κινδύνους. Τέταρτη τροπολογία, η υποχρέωση για τον ετούντα να διευκρινίζει εάν το αίτημα εξουδότησής του αφορά ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση ή μόνο ορισμένα κράτη-μέλη. Αυτό σε καμία περίπτωση δεν υποχρεώνει όλα τα κράτη-μέλη να ανταποκριθούν σε αυτό το έτοιμο. Ορισμένα κράτη-μέλη όπως η Γαλλία θα απαντούν πάντα αρνητικά. Πέμπτη τροπολογία, η υπενθύμηση της παιδιότητας ε, της αρχής της ε, προφύλαξης που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη σε αυτό το τομέα και στην εφαρμογή του. Είναι σημαντικό να το υπενθυμίσουμε. Αυτά κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρία εισηγητρία. Αυτές είναι οι παρατηρήσεις που επιθυμούσα να κάνω ως σκιώδης συζήτης. Ευχαριστούμε. Το λόγο τώρα έχει η συναλφούς Γκίλινγκ. Σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ απογοητεύτηκα, μάλλον, με τις τροπολογίες της κυρίας Ρίς για πολλούς λόγους. Αλλά, κυρίως επειδή εμένει σταθερά στην ε, στάση του Κοινοβουλίου που δεν ήταν πάντα ιδιαίτερο συνεκτική, όπως συχνά γίνεται στην πρώτη ανάγνωση με όλε αυτές τις τροπολογίε που περνάνε, ε, μένοντα λοιπόν ε, αμετακίνητα στις ε, τροπολογίες αυτές και ουσιαστικά επανακαταθέτοντας τις ίδιες τροπολογίες, παραμένει πολύ δύσκολη και πολύπλοκη αυτή η πρόταση και ουσιαστικά περιπλέκεται και παραπάνω αν προσθέσουμε και τα θέματα επισήμανσης. Το θέμα είναι κατά πόσο θα επιτρέψουμε ή όχι στα κρατημέλη να λαμβάνουν αποφάσεις βάσει και άλλων παραγόντων πέραν από την ασφάλεια της υγείας και του περιβάλλοντος. Και για να πάμε και παραπέρα. Θεωρώ ότι διακυβεύεται έτσι η αρχή του να μην περάσουμε το πρόσκομα του Συμβουλίου σε ό,τι αφορά την αλλαγή της νομικής ε, βάσης. Για παράδειγμα, ε, εκ νέου κατατέθηκε αυτή η τροπολογία. Είναι αρκετά σαφές ότι η στάση του Συμβουλίου θα πρέπει να, θα πρέπει να παραμείνει ως νομική βάση η ενιαία αγορά, όπως πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και ουσιαστικά μεγάλο τμήμα της νομοθεσίας που συζητάμε εδώ πέρα που έχει προφανώς τεράστια ωφέλη για το περιβάλλον, γίνεται βάση της νομικής βάσης για την ενιαία αγορά. Για παράδειγμα, σε ό,τι αφορά τι πλαστικές σακούλε, θα τις συζητήσουμε αύριο. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Είναι ωφέλιμο, θεωρώ, να χρησιμοποιείται αυτή η νομική βάση. Γιατί επιμένει λοιπόν η κυρία Ρή με την ε, τοποθέτηση του Κοινοβουλίου να αλλάξει η νομική βάση, γιατί θεωρώ χωρίς να κρίνω και να επικρίνω τον σκοπό της νομοθεσίας, την βολεύει η νομική βάση που έχουμε αυτή τη στιγμή. Γιατί οι ανησυχίες για τον ανθρώπινο οργανισμό και τις επιπτώσεις στον ανθρώπινο οργανισμό υπήρχαν ήδη σε κοινωτικό επίπεδο και αυτό αποτυπώνεται σε επίπεδο νομοθεσίας. Η νομοθεσία αυτή δεν έχει αυτό το σκοπό και αν το Κοινοβούλιο ε, επιμείνει στις θέσεις του δεν θα περάσει τίποτα τελικά από πλευράς νομοθεσίας σε ό,τι αφορά την απαγόρευση βάση περιβαλλοντικών παραγόντων, σε ό,τι αφορά την ε, ανθεκτικότητα σε γάματα ομικρών. Αυτά υφίστανται ήδη και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε επιχειρήματα αναδρομικά. Γιατί πολύ απλά αυτό ε, γελιοποιεί την ε, διαδικασία έγκρισης της ΕΦΣΑ. Μετά από όλα αυτά, στην πρώτη ανάγνωση είχα την αίσθηση, να σας πω την αλήθεια, ότι ήταν μια ακατάλληλη ε, απόπειρα από πλευρά του Κοινοβουλίου και δεν την υποστηρίξα. προσθέτονται, τόσο πολλά καινούργια σημεία που τελικά χάνουμε κάθε νομική βεβαιότητα. Αν συνεχίσουμε όμως αυτή τη διαδικασία θεωρώ ότι θα υπάρχουν και άλλοι τομείς που θα πρέπει να βελτιώσουμε και θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι τα μέτρα με παρεμποδίζουν τη σχετική έρευνα. Πολλοί φαίνεται εδώ πέρα στην αίθουσα να πιστεύουν ότι Υπάρχει μια τεράστια, ένα τεράστιο κίνημα που προσπαθεί να επιβάλλει τους γάματα ομικρών στην Ευρώπη. Δεν είμαι ενήμερη για κάτι τέτοιο. Αυτό που θέλει η βιομηχανία είναι να συνεχίσει η έρευνα. Και νομίζω ότι θα ήταν πάρα πολύ κρίμα αν με την νομοθεσία αυτή ε, ανακηρύσαμε παράνομη την έρευνα για τους γάματα ομικρών. Θεωρώ ότι θα πρέπει να προστατεύσουμε την έρευνα στα πλαίσια της κοινωνίας και των επιχειρήσεων. Επίσης θα πρέπει να κοιτάξουμε τα θέματα που αφορούν τους σπόρους, το οποίο βέβαια κοιτάξαμε, προστασία των καταναλωτών και των αγροτών σε ό,τι αφορά την ενιαία αγορά και διεθνείς υποχρεώσεις της Ένωσης. Αυτά είναι θέματα που θα θίξω στις τροπολογίες μου. Αλλά θα επανέλθω στο βασικό μου σημείο. Αν θέλετε πραγματικά να δώσετε στα κράτη-μέλη κάποιο περιθώριο απόφασης προκειμένου να μπορούν να λένε ότι δεν θέλουμε στην επικράτειά μας τέτοια καλλιέργεια, θα πρέπει να παραμείνει απλή η διαδικασία. Αν χρησιμοποιήσετε τη δικαιολογία αυτή για να λύσετε και άλλα προβλήματα, πολλά πολλά κράτη-μέλη το κάνουν, ουσιαστικά έχουμε χαράξει τον δρόμο της αποτυχίας. Ευχαριστούμε πολύ. Το λόγο έχει συνάδελφος Μπόιλεν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε την κυρία Ρή. και έφερε βελτιώσεις στο αρχικό σχέδιο κειμένου. Πρώτα-πρώτα έχουμε και την αλλαγή της ε, νομικής βάσης. Από το, το κομμάτι που αφορά την ε, στο Αγορά πήγαμε στο 192 που αφορά το περιβάλλον. Έτσι, με αυτό το νομοθέτημα τα κρατη μπορούν να αποφασίσουν εάν θέλουν γάμματα φόντου στην επικρατεία τους. Γι' αυτό και αν δεν είχαμε το 192 θα ήταν παράδοξη επιλογή η διάταξη που αφορά την εσωτερική αγορά. Να δούμε τι θα γίνει όσον αφορά την αδειοδότηση. Θα πρέπει με αυτή την νομοθεσία να μπορούν τα κρατημέλη με παράλληλα μέτρα να εξασφαλίσουν ότι τα γειτονικά τους κρατημέλη επίσης δεν έχουν γάμα ταφ όμικρον. Εν πάση περιπτώσει θα πρέπει ένα κράτο, να μπορεί να αποφασίσει αν θα έχει ή όχι γάμα ταφ όμικρον στην επικρατεία του. Είπαμε εδώ με ποια αιτιολογικά ε, μπορεί το κρατός μέλος να δώσει να μην δώσει την αδειοδότηση. Πάντως αυτά τα κριτήρια είναι πολύ περιοριστικά. Δεν δίνουν στα κράτη-μέλη το αναγκαίο περιθώριο για να μπορούν να κρίνουν αν θα απαγορεύσουν ή όχι την καλλιέργεια των οργανισμών αυτών. Επίσης, βλέπω ότι η κυρία Ρίες έχει τις τροπολογίες 22 και 24 για να βελτιώσει τη διαδικασία, αλλά θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει με το αν υπάρξουν έτσι προηγούμενα. Οπότε νομίζω ότι θα πρέπει σχετική παράγραφος που δεν είναι καθόλου ικανοποιητική για μια δημοκρατική κυβέρνηση θα πρέπει να διαγραφεί. Δεν είναι δυνατόν ένα κυριακό κράτος να ζητεί την άδεια από κάποιους βιομηχάνους για το αν θα επιτρέψει την καλλιέργεια αυτών των οργανισμών. Ευχαριστούμε, λέει ο Πρόεδρος. Ο κύριο Στάσ πάλι, ζητώ το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε και συνάδελφοι. Πρέπει να ομολογήσω ότι είμαι αρκετά ικανοποιημένο ε, από τη συνεργασία με τους συζητητέ και με τους κοιότε. Δύο φορέ συναντηθήκαμε, διαβουλευτήκαμε και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και με την Προεδρία. Αλλά, καταρχάς, πριν από κάθε συζήτηση για το θέμα αυτό, θα ήθελα να υπογραμμίσω το γεγονός ότι ο πρόεδρος, ο μοναδικός πρόεδρος Γιούγκερ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έκανε σημαντικές δηλώσεις σε ό,τι αφορά τους γαματάφ ομικρών στην ομιλία του προς το Κοινοβούλιο και προς τις μεμονωμένες πολιτικές ομάδες και στην, στο Mission Statement, στην ε, επιστολή προ τον Επίτροπο Αντρεκάιτης δεσμεύθηκε ότι μετά από έξι μήνες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα υποβάλει καινούργιες προτάσεις. Νομίζω λοιπόν ότι είναι επίγον το θέμα και θα πρέπει να διεξαχθεί τριμερής διάλογος και με το Συμβούλιο για να ξέρουμε τι ξεκινάμε και προς τα ποια κατεύθυνση θα κινηθούμε. Δεν ε, συζητάμε χωρίς να ξέρουμε ποιες είναι οι συγκεκριμένες προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δεύτερο στοιχείο. Χαίρομαι που η συγγήτρια στην έκτασή της καταθέτει πολλές τροπολογίες για τις οποίες αγωνιστήκαμε στην πρώτη ανάγνωση με την κυρία Ρεπάζ, την προκάτοχό της. Και ιδιαίτερος με ικανοποιεί η αλλαγή της νομικής βάσης. Κάναμε συζήτηση με την Ιταλική Προεδρία σχετικά με το θέμα αυτό και με την νομική υπηρεσία του Συμβουλίου και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχω πιστεί στην παρούσα φάση. Υποστηρίζει λοιπόν την εισηγήτρια σε ό,τι αφορά την αλλαγή της νομικής βάσης. Και χαίρομαι ιδιαίτερος με την αναφορά που κάνει η εισηγήτρια στην εκτέλεση των ε, συμπερασμάτων ε, του Συμβουλίου του Δεκεμβρίου του 2008 και σε ό,τι αφορά τις κατευθύνες γραμμές για τους γάμματα όμικρων που δεν μπορούν να βασίζονται μόνο σε θέματα ισοτιμίας, αλλά θα πρέπει να εξετάζονται οι άμεσες και έμεσες συνέπειες και τα επιστημονικά στοιχεία. Τροπολογία βαριθμών 3 της Και χαίρομαι ιδιαίτερως με διάφορες ε, τροπολογίες που καλούν για περισσότερη διαφάνεια, δημοσίευση των κοινοποιήσεων, των αποφάσεων, των ε, συμφωνιών. Η απόλυτη διαφάνεια θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντική και εδώ περνάμε στα πιο δύσκολα. Η πρόταση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για να υπάρχει ένα σύστημα διφασικό, δύο φάσεων. Το είπε και η κυρία Μπόιλεν, το γεγονός ότι στην πρώτη φάση ουσιαστικά δίδεται λέγειν στους παραγωγούς γαμάτα όμικρον στην πρώτη φάση για την τελική λήψη απόφαση είναι κάτι απαράδεκτο πραγματικά για μας τους πράσινους. Γι' αυτό λοιπόν και θα καταθέσουμε τροπολογίες προκειμένου η πρόταση του Συμβουλίου για την πρώτη και την δεύτερη φάση να ακυρωθεί. Να προσπαθήσουμε να ακυρωθεί. Και να εργαστούμε Προ την κατεύθυνση τη δεύτερη φάση, αυτό που ονομάζεται τώρα δεύτερη φάση. Και στην δεύτερη ανάγνωση λοιπόν το Κοινοβούλιο θα πρέπει να ορίσει υγιή νομικά κριτήρια προκειμένου τα κράτη-μέλη να έχουν την ευκαιρία να λάβουν τις αποφάσεις που θέλουν να λάβουν με πλήρη ανεξαρτησία και σίγουρα σε καμία περίπτωση μέσω επαφών ή οποιασδήποτε παρέμβαση των παραγωγών γάματα αφόμικρων οι οποίοι ενδεχομένω να επηρεάσουν την τελική λήψη αποφάσεων. Γι' αυτό και είναι πάρα πολύ σημαντική η τροπολογία υπαριθμών 24 για μια μη δεσμευτική, μη εξαντλητική λίστα των λόγων απαγόρευσης. Συμπεριλαμβάνει βλέπω η συγγήτρια τη λίστα που είχαμε συμφωνήσει με την κυρία Λεπά, στην οποία είχε υποστηρίξει μεγάλη πλειοψηφία. Το τονίζω αυτό στην πρώτη ανάγνωση. Είναι σαφές το πολιτικό μήνυμα. Και καλό τους συναδέλφους, θα τους ε, μιλήσω και προσωπικά. Όσοι έχουν αμφιβολίες ε, για την πρώτη φάση, μήπως θα μπορούσαμε από μαζί να καταθέσουμε τροπολογίες για να ακυρωθεί, να καταργηθεί αυτή η πρώτη φάση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Κλείνουμε το κύκλο των ε, σχεδόν εισηγητών και δίνουμε το λόγο στη συναλφέρη. Εύη. Λοιπόν, και εμείς θα θέλαμε να υπογραμμίσουμε βάση του άρθρου 192 μπορεί να δημιουργηθεί πρόβλημα με το αναφέρεται στο 26β στην παραγραφό 3 όπου προβλέπει η δυνατότητα προσφυγής σε αιτίες κοινωνικο-οικονομικές ή χωροταξίας που δεν μπορούν να αιτιολογηθούν με θέματα περιβαλλοντικά όπως θα ήθελε η νομική βάση προτείνουμε ενδεχομένως να εισαγούμε και τις δύο νομικές βάσεις για πιο μεγάλη ευελιξία. Παρά τις προσπάθειες της ηγήτριας, την οποία ευχαριστούμε για τη δουλειά της, ε, παρόλα αυτά η δυνατότητα ένας ιδιώτης να μπορεί να αρνηθεί ένα αίτημα ενός κράτους μέλους μας φαίνεται απαράδεκτο. Το πρόβλημα είναι καθαρά πολιτικό. Δεν υπάρχουν άλλες ε, διατυπώσεις παραδεκτές. Πρέπει να διαγράψουμε τη διαδικασία. Αλλιώς θα ήταν σαν να ε, παρα, παρατάμε την κυριαρχία ενός κράτους μέλους, αν δεν καταλείπουμε. Όσον αφορά την τροπολογία 27, η πρόταση που υπάρχει στην παραγραφό 5β, η απαγόρευση να βασίζεται σε κάποια ανάλυση κόστος που να περιέχει και πιθανές εναλλακτικέ, δεν φαίνεται να έχει συνοχή με τη διευκόλυνση των διαδικασιών λήψη απόφαση στα κράτη-μέλη όσον αφορά την καλλιέργεια των γενετικώς οργανισμών. Εμεί θεωρούμε λοιπόν ότι αυτό βάζει περισσότερα εμπόδια. Τέλο, θέλαμε να υπογραμμίσουμε ότι η εισαγωγή τη υποχρεωτική φύση των σχεδίων συνύπαρξη θα μπορούσε να αποδυναμώσει την νομοθεσία από τη στιγμή που θα πρέπει να προσδιορίζονται οι συνθήκες υπό τις οποίες μπορούν να συνεπάρχουν ε, οι δύο καλλιέργειες ε, και μάλιστα μαζί με βιοδυναμικές ή βιολογικές καλλιέργειες. Αντιθέτως θα έπρεπε να αφήσουμε κάθε κράτος ε, μέλος ελεύθερο να υιοθετήσει τα σχέδια εφόσον αποφασίσει να δώσει το πράσινο φως για την καλλιέργεια γενετικώς τροποποιημένων φυτών. Ευχαριστούμε. Ας ξεκινήσουμε τώρα με τις παρεμβάσεις των υπολείπων συναδέλφων έχετε τρία λεπτά ώστε να μπορέσουμε να κλείσουμε έγκαιρα τη συζήτηση. Ξεκινάμε τη συναδελφή κυρία Πιλαραγιωσό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ την εισηγήτρια αλλά και τους κοιόδες και εισηγήτρια. Ναι. Πρώτα για περίπλοκο ζήτημα, το οποίο είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και συνεργαστικό. Να σας πω τις σκέψεις μου επί της ε, ουσίας. Ε, βέβαια είναι και το θέμα της νομικής βάσης οι γαμάτα φωνηρών τελικά αφορούν μια τεχνική βελτίωση των φυτών. Στην Αμερική αυτά έχουν ξεκινήσει εδώ και 40 χρόνια. Είχαμε τότε κάποιο είδους πιο αυθόρμητη επιλογή των καλύτερων φυτών και τελικά αυτό ήταν η μέθοδος. Όμως αυτό που θα πρέπει να γίνει εδώ είναι ότι θα πρέπει να ισχύσουν για τους γάμματα φαινομικρών τα ίδια όσα ισχύουν για την καλομεταχείριση των ζώων και για τα φυτοϊγειονομικά. Να ληφθεί υπόψη επομένω η ΕΦΣΑ, οι συναρμόδιες εθνικές αρχές και έτσι να λαμβάνονται οι αποφάσεις. Γι' αυτό και εγώ δεν συμφωνώ με κάποιες από τις τροπολογίες της συζυγήτριας που αμφισβητεί τέτοιου είδου ε, ισορροπία δυνάμει όσον αφορά της, ε, που είναι επιστημονική τεκμηρίωση για τις αποφάσεις. Οι επιστημονικές μελέτες δεν είναι κάτι που θα προσαρμόζεται ε, στα κέφια μας. Είναι δεδομένες. Μια χώρα ναι, μπορεί να μην θέλει να έχει στην επικρατειά της γάμματα Το κάθε κράτος να έχει την ευχέρεια να προβεί σε αυτή την επιλογή. Και δεν χρειάζονται προφάσεις και δικαιολογίες περιβαλλοντικές ή άλλες. Τόσον αφορά τις ε, τροπολογίες για την υποχρεωτικότητα, για τα μέτρα ε, της συνεπούς εφαρμογής και ομοιογενούς. νομίζω δεν είναι εδώ αυτή η οδηγία το νομοθέτημα που θα πρέπει αυτά να αναγραφούν. Δεν έχουμε ακόμα ολοκληρώσει τις σχετικές μελέτες. Δεν ξέρουμε ακόμα ε, πολλά για την κάθε ποικιλία, για το κάθε φυτό για την κάθε καλλιέργεια. Θα πρέπει κανείς να έχει μια σφαιρική γνώση των ε, επιστημονικών μελετών, τις λαμβάνει όλες υπόψη και να μπορεί να τις προσαρμόσει στα κέφια του για να τις χειραγωγήσει. κύριε Πρόεδρε. Ήθελα να πω για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο σημείο που θα πρέπει να δικαιολογήσουμε γιατί θέλουμε αυτή την τακτική, την συνήθεια διαδικασία και όχι την διαδικασία της συναπόφασης. Γιατί το Συμβούλιο θέλει εμείς να συναποφασίζουμε. Γιατί υπήρξε απόρριψη όλων των προτάσεων. Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή απεφάνθη σαφώς. Θεωρεί ότι η νομική βάση θα πρέπει να αλλάξει. Και παραλαμβάνομαι ότι είναι κάτι πολύ σημαντικό νομική βάση. Αυτό διαφέρει από το να πούμε επομένω ότι θέλουμε ε, την διάταξη για την ενιαία αγορά ως νομική βάση. Άλλωστε, η διακριτική ευχαίρεια των κρατών μέλων πιθέται ένα αμφιβόλο. Θέλουμε την προσέγγιση που αφορά τη διάταξη για το περιβάλλον, σαν νομική βάση. Και πολλοί λόγοι μας ε, οδηγούν σε αυτή την επιλογή. Στην πρώτη φάση είπαμε ότι θα πρέπει να ισχύσει κάτι τέτοιο αλλά δεν ξέρω γιατί η τροπολογία θα πρέπει να λέει ότι μόνο οι υπορισμένες περιστάσεις ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ε, κάνει τις ενέργειες που προβλέπει. Μα τι θα φιλτράρει δηλαδή την ε, αίτηση για διοδότηση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εγώ δεν βλέπω αυτό να δικαιολογείται. Νομίζω ότι δεν πρέπει τα κρατημέλη να στερούνται της διακριτικής ευκαιρίας και νομίζω ότι αξίζει συγχαρητηρίων η εισηγήτρια γιατί προσπάθησε να καταλήξει στον καλύτερο δυνατό συμβασμό. Εγώ προέρχομαι από ευρωσκεπτικιστικό κόμμα της Ουγγαρίας. Εμείς λέμε όχι στις τεχνικές σχετικές με τους γάματα φόμικρων. Και αυτό που κάνουμε τώρα προσπαθούμε να δώσουμε στα κράτη-μέλη όσο γίνεται ευρύτερο περιθώριο ελιγμών. Και λέμε ότι αν ένα κράτος πει όχι, όταν έχουμε μια ολόκληρη διαδικασία, ε, μια ολόκληρη ε, ε, διαβούλευση, γιατί μετά καταλήγει σε ένα ναι, σε ένα όχι. Μα είναι προνόμιο του κράτους μέλους να λαμβάνει αυτή την απόφαση. Για να μην έχουμε λοιπόν εμβαλωματική λύση. Λόγω συναδέλφο Ολβένη. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, το ζήτημα είναι εξαιρετικά περίπλοκο και πιστεύω ότι πρέπει να προσπαθήσουμε να εκφραστούμε απλά και σαφώς. Έχουμε μπροστά μας μια υπόθεση στην οποία προσπαθούμε να βρούμε μια λύση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. δεν μπορούμε να σκεφτόμαστε το ενδεχόμενο λύσεων ανακράτος μέλος για τέτοια ζητήματα. Εγώ πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό και ευχαριστώ την κυρία εισηγήτρια που έφτασε μέχρι αυτό το σημείο. Όλα τα επόμενα βήματα δεν πρέπει να θέσουν σε κίνδυνο τα αποτελέσματα που έχουμε επιτύχει μέχρι στιγμή. Γιατί ο κίνδυνο είναι ο εξή. Προσπαθούμε να τραβήξουμε λίγο τα ε, όρια και υπάρχει κίνδυνο ε, για ένα αποτέλεσμα εντελώ αβέβαιο. Διαδικασίες οι οποίες ε, θα είναι εξαιρετικά σύνθετες. Αν έχουμε ένα κράτος το οποίο θέλει να μην ε, δεχθεί στους γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς, πρέπει να μπορούμε να διασφαλίσουμε στο κράτος αυτό αυτή τη δυνατότητα. Εμείς έχουμε ήδη προωθήσει τέτοιες αποφάσεις και λάβει τέτοια μέτρα. Όσον αφορά τη διασυνοριακή μόλυνση, δεν πρέπει να υποτιμάμε το γεγονός ότι τέτοιες απαγορεύσεις ε, μειώνουν τέτοιου είδους μόλυνση. Πρέπει να λαμβάνονται τέτοια μέτρα. Και σε περίπτωση μόλυνση πρέπει να εφαρμόσουμε την αρχή ο ρηπαίνων πληρώνει. Αλλά είμαστε πολύ μακριά από όλα αυτά εγώ πιστεύω ότι η ΕΦΣΑ στην ανάλυση κινδύνων της πρέπει να μπορεί να διεξάγει η ΕΦΣΑ μια ανάλυση κινδύνων. Εκεί πιστεύω ότι πρέπει να κάνουμε μια τροποποίηση. Και για να μην ξεπεράσω το χρόνο μου θέλω να υπογραμμίσω κάτι τελευταίο. Όλοι, όλοι οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν το δικαίωμα να γνωρίζουν τι τρώνε, τι καταναλώνουν. Μπορούμε πιστεύω να βρούμε συμβιβασμούς, αλλά η βασική αρχή πρέπει να είναι αυτό το ανθρώπινο δικαίωμα το οποίο πρέπει να σεβαστούμε. Πιστεύω λοιπόν ότι στην νομοθεσία δεν πρέπει να ξεχνάμε νομοθετώντας αυτή τη θεμελιώδη αρχή. Ευχαριστούμε πολύ. Το λόγο έχει ο συνάδελφος κύριος Όσλινγκ. να σας πω κάτι το οποίο θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε όταν μιλούμε για την απαγόρευση από πλευρά κράτου μέλους θα πρέπει να μην ξεχνούμε το ότι υποσχέθηκε ο κύριος ε, Γιούγκερ μια διαδικασία διοδότηση ω τμήμα της όλης υπόθεσης. Οπότε όλα αυτά θα συζητηθούν το επόμενο εξάμεινο από κοινού. Δεν μου αρέσει η ισχύουσα διαδικασία. Δεν είναι δημοκρατική. Λέει ο κ. Χάσλιν. Τα κριτήρια της ΕΦΣΑ δεν είναι για όλους σαφή. Δεν είναι κατανοητά. Επομένως και αυτά θα αποτελέσουν αντικείμενο ε, διαπραγμάτευσης. Εγώ αυτό φοβάμαι. Ότι θα έχουμε τελικά απαγορεύσεις και deal που θα κλείνουν τα κράτη-μέλη με μεγάλες εταιρείες. για τα τροποποιημένα όσον αφορά την επικρατεία τους. Με ευρωπαϊκή αδειοδότηση θα έχουμε ενιαίο σύστημα για όλη την Ευρώπη. Αυτό τι σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχουν δεσμευτικοί κανόνες. Δεν είναι δυνατόν... Θα πρέπει να υπάρχουν αποστάσεις από τους ε, από τη βιολογική καλλιέργεια, για παράδειγμα, και σε ό,τι αφορά τη διαφάνεια. Θα πρέπει να υπάρχει διαφάνεια προκειμένου όλοι να ξέρουν τι γίνεται σε κάθε έκταση. Πού καλλιεργούνται γάμα, ταφ, ομικρον. Όλα αυτά λοιπόν συγκαταλέγονται στο πακέτο. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να υπάρχουν συγκεκριμένα δικαιώματα σε κάποια κρατημέλη, τα οποία δεν υπάρχουν σε άλλα κρατημέλη και σε ό,τι αφορά τους ε, παραγωγούς και τους καταναλωτές. Χρειαζόμαστε λοιπόν ευρωπαϊκούς κανόνες, πιο αυστηρούς κανόνες και θα πρέπει να αλλάξουν σχετικές διαδικασίες. Σε κάθε περίπτωση τον κύριο Γιούγκερ ε, θα του υπενθυμίσουμε όλα όσα μας υποσχέθηκε. Ευχαριστούμε πολύ, ε, συνάδελφος κυρία Πέτερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω μόνο το εξή. Στην Κροατία δεν επιτρέπεται η διάθεση στην αγορά ζώνων, γάμα ταφ όμικρον. Αλλά οι μέλισσες, ο άνεμος, δεν γνωρίζει προς τα πού πάμε και πού υπάρχουν γάματα αφόμικρον. Άρα λοιπόν θα πρέπει να συμπεριληφθεί άλλο ένα στοιχείο. Ε, το στοιχείο των μέτρων πρόληψης σε ό,τι αφορά και το σχετικό πρωτόκολλο. Αυτό δεν σημαίνει ότι η δημόσια γνώμη μετά τη συνθήκη του όρχους θα πρέπει να συμμετέχει Πρέπει να σας πω ότι ανησυχώ ιδιαίτερως ότι αφορά την πρόταση που έχουμε μπροστά μας. Γιατί η πρόταση αυτή θα σήμαινε ότι μετά από την αξιολόγηση κινδύνου της σχετικής ε, επιτροπής δεν θα χρειαστεί να αποδεικνύεται ότι δεν υπάρχουν αρνητικές επιπτώσεις ε, των ενδεχόμενων προϊόντων Αντιθέτως, ότι τα κρατημέλη θα πρέπει να αποδεικνύουν ότι υπάρχει κίνδυνος για να υπάρχει οποιοδήποτε περιορισμός για την καλλιέργεια γάμματα αφόμικρων. Οι πολίτες δε στα κρατημέλη έχουν διαφορετικές δυνατότητες προστασίας. Δεν προστατεύονται με τον ίδιο τρόπο και γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει γίνεται δυνατή η διαδικασία διαβούλευσης διασυνοριακά. Αυτό είναι κάτι εντελώ καινούριο ό,τι αφορά την προστασία του περιβάλλοντος στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ελπίζω ιδιαίτερω στο μέλλον να μην υπάρξουν, να μην χρειαστεί πουθενά άλλου αλλαγή νομοθετική πράξη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε λοιπόν να προχωρήσει σε μια τέτοια καθολική ρύθμιση. Θα ήθελα να ευχαριστήσω σε όσους αναφέρθηκαν στην αλλαγή της νομικής βάσης από το 114 στο 129 και θα ήθελα να ευχαριστήσω σε όσους υπέδειξαν τη λανθασμένη λογική που κρύβεται πίσω από την αλλαγή αυτή. Δεν μου βοηθάει να αντιμετωπίζουμε ένα κυρίαρχο κράτο σαν ανεπιχείρηση. Δεν είναι ούτε ωφέλιμο ούτε ευκταίο αυτό. Γι' αυτό λοιπόν αυτό επιθυμώ να αλλάξει. Ευχαριστώ πολύ. Thank you. I'm going to continue to chairing. Ο πρόεδρος. Εγώ θα συνεχίσω να προεδρεύω. Ο κ. Μαζουρόνης είναι ο επόμενος αγορητής. Λίγο να πληρωτήσω του πρόεδρου. Αγαπητοί συνάδελφοι, οι μακροπρόθεσμες επιπτώσεις των ε, τροποποιημένων για τον άνθρωπο δεν έχουν ακόμα διερευνηθεί πλήρως, άρα θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί να μην βιαζόμαστε. Θα πρέπει να ξέρουμε ακριβώς υπό ποιες συνθήκες θα προστατεύεται και το περιβάλλον σου γίνεται περισσότερο γιατί είναι χωρίς επιστροφή οι συνέπειες από τα τροποποιημένα. Προσοχή επομένως, ασφάλεια, ούτω ώστε να υπάρχει προπαρασκευή, προετοιμασία κάποιων μηχανισμών προστασίας. Να έχουμε κάποιο ανοιχτό κατάλογο με τα σχετικά κριτήρια. Άρα, εάν θέλουμε ασφάλεια δικαίου, τότε θα πρέπει να εξασφαλίσουμε αυτούς τους 24 μήνες για να υπάρξει μεταφορά στο δίκαιο των μελών των όσων επιβάλλονται. Να ετοιμαστούν τα κρατημέλη και το δίκαιό τους. Οι έξι μήνες δεν φτάνουν. Επίσης για την κοινοποίηση πάμε στους 12. Άρα να δούμε τι γίνεται με τις προθεσμίες αλλά και με τους χωρισμούς. Δεν γνωρίζουμε επί ποιας βάσεως ε, προτάθηκαν τα δύο χρόνια ούτως ώστε το κρατός μέλος να μπορεί να ζητήσει κατάργηση της ε, περιοχής που θα αφορά τους γαματαφόμικρους. θα πρέπει να μπορεί κανείς να αντιμετωπίσει κάθε αλλαγή στις νομικές ρυθμίσεις. Έχουμε επίσης αυτή την προθεσμία των 75 ημερών, μέσα στις οποίες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να ερευνήσει τα σχετικά με αίτηση από κράτους μέλους. Προσοχή μην έχουμε εδώ πέρα παραθυράκια στον νόμο. Και να νομιμοποιούνται τα τροποποιημένα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά όχι σε εθνικό επίπεδο. Γιατί έτσι είναι ανεφάρμοστη η ρύθμιση. Είναι σημαντικό τα κράτη-μέλη να είναι σε θέση να μπορούν να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα το συντομότερο. Και για τη Λιθουανία είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει ε, μια ανοιχτή λίστα κριτηρίων και διαχειριστές του κινδύνου να είναι τα κράτη-μέλη και αναλόγως να απαντούν στις αιτήσει για τα τροβημένα. Και χρειάζονται όλοι και δικαιώματα και περιθώριο ούτως ώστε να μπορούν να αποφασίσουν για το τι γίνεται με τα τροβημένα στην επικράτειά τους. Ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ και την κυρία Ρίση που είναι η συγγήτρια σε ό,τι αφορά την επικουρικότητα. Αυτό θα πρέπει να είναι η βασική αρχή. Θα πρέπει η ευθύνη να παραμένει στα χέρια της, του κράτους μέλους και μας ικανοποιούν οι τροπολογίες της συγγήτριας. Αλλά αυτό δεν θα πρέπει να σημαίνει αβεβαιότητα για τους παραγωγούς και τους καλλιεργητές. Αλλά να μην ξεχνάμε και τον καταναλωτή, τον πολίτη. Η συγγήτρια λαμβάνει υπόψη τα θέματα στα διασυνοριακά και τους κινδύνους που ενέχονται. Λαμβάνεται υπόψη η μεταβατική φάση για τους ε, ε γεωργούς που καλλιεργούν γάμα τα όμικρον, αλλά αν συμπεριληφθεί η υποχρέωση έρευνας για εναλλακτικέ, θα πρέπει να είναι σαφές ποιος θα έχει την ευθύνη για το θέμα αυτό. Και το πιο σημαντικό σημείο από δική μου πλευρά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να μπορεί η ίδια να αποφασίσει να δώσει νομικό κύρος στην καθεστώς στις απόφασεις της ΕΦΣΑ γιατί είναι πολύ κατηγορηματική η τετραετής περίοδος που διευκρινίζεται. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ένα εκτελεστικό όργανο και θα πρέπει λοιπόν να μπορούμε εμείς να εξετάζουμε ε, και με το δικό μας ρυθμό να δίνουμε έγκριση. Αυτό σε ό,τι αφορά τις κατευθυντήριες γραμμές, σε ό,τι αφορά το περιβάλλον και την προστασία του περιβάλλοντος. Η αρχική στάση του Συμβουλίου μου φαίνεται καλύτερη και θα ήθελα να ακούσω τι έχει να απαντήσει η ή άλλο θα καταθέσω σχετική τροπολογία. Ευχαριστώ. Το επόμενο σχόλιο θα το κάνω εγώ και θα μιλήσω στα ουγγρικά. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια την κυρία Ρης ε, για τη δουλειά που έχει κάνει. Οι τροπολογίες ε, που παρουσιάζει βελτιώνουν σε μεγάλο βαθμό την αρχική πρόταση και απαντούν ε, σε πολλά προβληματικά σημεία. Ήθελα να επιστήσω την προσοχή στο εξή. Χαίρομαι που αναφέρεται η διασυνοριακή μόλυνση στις τροπολογίες και η υποχρέωση των κρατών μελών να ληφθούν μέτρα. Είναι θεμελιώδης σημασία διότι ένα κράτος μέλος για να μην έχει γενετικό τροποποιημένου οργανισμούς καθόλου πρέπει να εφαρμόσει προστατευτικά μέτρα ώστε να αποφευθεί διασυνοριακή μόλυνση. Ωστόσο, πρέπει να αναγνωρίσουμε το γεγονό ότι το ζήτημα αυτό δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί σε εθνικό επίπεδο μόνο. Εάν αναθέσουμε το καθήκον αυτό στα κράτη-μέλη μόνο, κάθε κρατός μέλος ε, θα έπρεπε να έχει διαφορετικά μέτρα προστασίας ε, εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα βρεθούμε σε μια παράδοξη κατάσταση όπου μπορεί ένα κράτος ε, να έχει διαφορετικά μέτρα από τη μία πλευρά των συνόρων και από την άλλη πλευρά των συνόρων να υπάρχουν άλλα μέτρα σε αυτές τις γειτονικέ περιοχές. Γι' αυτό το λόγο είναι σημαντικό για να επιτευχθεί ο στόχος αυτής της καταταλάριστες τροπολογίες, να υπάρχουν ελάχιστα κριτήρια σε ευρωπαϊκό επίπεδο τα οποία θα ρυθμίζουν τις ελάχιστες απαιτήσει που θα δίνουν τη δυνατότητα ένα κράτος μέλος να είναι απαλλαγμένο από τους γενικούς οργανισμού οργανισμούς εφόσον έχει αποφασίσει την απαγορεύσή τους και να μην ε, βρίσκεται σε μια κατάσταση όπου έχει κάποιο σύστημα μη διαφανές το οποίο δεν είναι διαχειρίσιμο ούτε νομικά. Εγώ θα υποβάλω τροπολογίες προς αυτή την κατεύθυνση. Θα ήθελα σε κάθε περίπτωση να επιστήσω την προσοχή των συναδελφών σε αυτό το σημείο το οποίο θεωρώ εξαιρετικά σημαντικό και πρέπει να απαντήσουμε. Ο τελευταίος ομιλητή είναι ο κύριο Τζαρντίνη. Η κυρία Τζαρντίνη, συγγνώμη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι γρήγορη, τα περισσότερα έχουν ήδη υποθεί. Συμμερίζομαι και εγώ και ευχαριστώ την εισηγήτρια για το έργο της. Συμμερίζομαι στις βασικές ιδέες παρότι έχω και ψεπιφυλάξεις επιφυλάξεις και τις που έχω εκφράσει ήδη. Σίγουρα πρόκειται για μια συζήτηση δημοσίου ενδιαφέροντος με πολλές αντιφάσεις ε, και γενικά η κοινή γνώμη είναι αντίθετη. Και γενικά υπάρχει ένα πρόβλημα συνύπαρξης μεταξύ των παραδοσιακών καλλιεργειών και των γενετικά τροποιημένων. Ο κίνδυνος ε, μόλυνσης πρέπει να διατηρηθεί υπό έλεγχο απολύτως. μια περιοχή στη Βορεια Ιταλία πριν κάποιο καιρό υπήρξε μια περίπτωση μόλυνσης DNA που είχε μεταφερθεί με τον αέρα και με τη γύρι και διαπιστώθηκε ότι στη γειτονική περιοχή η μόλυνση είχε φτάσει το 10%. Κατά την απόψή μας, εάν οι κανόνες ε, δεν είναι αυστηροί, υπάρχει η περίπτωση η μόλυνση να φτάσει σε σημείο τέτοιο σε μερικά χρόνια να οδηγεί σε πλήρη εξαφάνιση των παραδοσιακών καλλιεργειών. Και μετά θα πρέπει να βάλουμε την επισήμανση Γενετικός τροποποιημένων προϊόντων σε όλα τα προϊόντα γιατί σύμφωνα με την νομοθεσία μας αρκεί 0,9% για να θεωρηθεί ένα προϊόν γενετικώς τροποποιημένο. Τα μέτρα λοιπόν συνύπαρξης πρέπει να είναι αποτελεσματικά, θα πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα τη διασυνοριακή μόλυνση. Εγώ θεωρώ ότι για μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου μάλιστα θα πρέπει να Υπάρχει και ένας πιο λεπτομερής κατάλογος ε, αιτιών. Δεν είμαι βέβαιη, έχω κάποιες αμφιβολίες ε, για την περίπτωση των ε, ιδιωτικών συμφερόντων, γιατί δεν ξέρω κατά πόσο πρέπει να συμπεριληφθεί αυτό για να διασφαλίσουμε το δημόσιο συμφέρον. Θα υποβάλω λοιπόν σχετικέ τροπολογίες. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Φτάνουμε στο τέλος της οροσχολιασμού των μελών της Επιτροπής. Και τώρα το λόγο έχει η Κομισιόν από την πρόσφατη της DG Sanko για να απαντήσει στα διάφορα ερωτήματα. Merci, le Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να επιμείνω σε τρία σημεία. Πρώτα απ' όλα, οι δηλώσει του μελλοντικού Προέδρου, του κ. Γιούνκερ, στο επιστολή που απευθύνεται στον ε, επίτροπό μας ο κ. Γιουνκέρ ε, ανέφερε ότι θέλει εντός έξι μηνών να αναθεωρηθεί η διαδικασία λήψη αποφάσεων που αφορά την ε, άδεια καλλιέργειας και χρήσης γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών τόσο για καλλιέργειες όσο και για τη διατροφή ανθρώπων και ζώων. Ο μέλλον ε, επιτροπός μας, ο κύριος ε, Γιονικαίτης, θα πρέπει να αναλάβει αυτή την, ε, αυτό το καθήκον μέσα στο επόμενο εξάμενο και θα χρειαστεί να συζητηθεί. Είναι σαφές, κατά την απόψή μας, για την παλιά και τη μελλοντική Κομισιόν ότι αυτή η διαδικασία που έχουμε μπροστά μας και που αφορά την καλλιέργεια των γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών και τη δυνατότητα ενός κρατού μέλους να αρνηθεί, να απορρίψει τις καλλιέργειες αυτές στην επικράτειά του ανήκει σε μια από αυτές τις νέες ε, φιλοσοφίες, ιδεολογίες παρότι το είχαμε προτείνει από το 2010 χωρίς να γνωρίζουμε φυσικά τότε τις οδηγίες του μέλλοντος Προέδρου του κ. Γιούνκερ νομική βάση Τώρα θα χρησιμοποιήσουμε το 114 άρθρο το 192. Εμείς προτείνουμε το 114 γιατί... γιατί εκεί βασίζεται η οδηγία. Θεωρούμε ότι αυτό το άρθρο 114, αντίθετα με το άρθρο 192, προστατεύει όχι μόνο το περιβάλλον, όπως το άρθρο 192, αλλά προστατεύει το άρθρο 114 και την υγεία των ζώων, την υγεία των φυτών και την υγεία των ανθρώπων. Ενώ το 192 αφορά πολύ συγκεκριμένα το περιβάλλον. Γι' αυτό το λόγο θεωρούμε ότι το άρθρο 114 είναι προτιμότερο ως νομική βάση για την πρόταση αυτή η οποία τροποποιεί όπως γνωρίζετε το κομμάτι ενός άρθρου. Το τρίτο στοιχείο σε αυτή τη φάση 1 αφορά αυτή τη φάση 1 που είναι ε, κάτι που αμφισβητήσιμο. Δεν υπήρχε στην αρχική πρόταση της Κομισιόν, εισήχθη στη συνέχεια από το Συμβούλιο. Δεν ξέρω αν θα δώσετε το λόγο στην εκπρόσωπο του Συμβουλίου. Εμείς θεωρήσαμε ότι αποτέλεσε κάποια βελτίωση σχέση με τη φάση 2. επειδή θεωρούμε ότι δίνει περισσότερη εξουσία και περισσότερες ελευθερίες στα κράτη-μέλη. Ουσιαστικά δίνει λιγότερα δικαιώματα στις ε, επιχειρήσεις γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών. Δίνει πολύ μεγαλύτερη εξουσία και ελευθερία στα κράτη-μέλη, τα οποία μπορούν να αποφασίσουν, χωρίς να το αιτιολογήσουν, να αποφασίσουν λοιπόν να ζητήσουν από μια επιχείρηση να μην καλλιεργήσει γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς στην επικράτειά τους. Διότι όπω έχουν τα πράγματα αυτή τη στιγμή, μια εταιρεία γενετικώ τροποποιημένων ε, οργανισμών ζητά άδεια καλλιέργεια ε, και στα 28 κράτη-μέλη. Εάν διατηρηθεί λοιπόν αυτό το βήμα, το κράτος μέλος θα έχει το δικαίωμα να ζητήσει να μην γίνουν καλλιέργεια στην επικρατεία του. Ε, θεωρούμε λοιπόν ειλικρινά ότι αυτή η φάση 1, αυτό το βήμα 1, παρέχει περισσότερες εγγύσεις στο κράτος μέλος. Του παρέχει τις νομικές εγγύσεις ώστε να μπορεί να αρνηθεί καλλιέργεια τέτοια στην επικρατεία του, το οποίο δεν συμβαίνει σήμερα. Ορισμένα κρατημέλη έχουν νομοθετήσει εθνικά την απαγόρευση των καλλιεργειών, αλλά όπως γνωρίζουμε όλοι, αυτές είναι αποφάσεις που νομικά είναι λίγο ευάλωτες και μάλιστα αντίκεινται στο κοινοτικό δίκαιο. Γι' αυτό το λόγο, παρότι εμείς, ε, δεν ήμασταν εμείς που επινοήσαμε αυτό τη φάση 1, θεωρούμε ότι επιφέρει κάποιες βελτιώσεις στην αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε, φυσικά θεωρούμε επίσης ότι πρέπει να σχετίζεται με τη φάση 2, δηλαδή ότι πρέπει να ξεκινάμε με τη φάση 1 πριν ξεκινήσουμε τη φάση 2. Αυτά είναι συντομία τα τρία βασικά σημεία που ήθελα να αναπτύξω εδώ. Τώρα το θέμα που αφορά την αιτιολόγηση και τη διεύρυνση της ε, λίστας ε, αιτιολογήσεων. Σήμερα έχουμε 7 που περιλαμβάνουν τις αιτίες που είχε προτείνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά την πρώτη ανάγνωση. Χρειάζονται διευκρίνηση, χρειάζονται επεξηγήσει, χρειάζονται περισσότερη ανάλυση, πιο λεπτομερή περιγραφή. Εμείς θεωρούμε ότι όσο περισσότερες λεπτομέρειες υπάρχουν, τόσο πιο περιοριστικά γίνονται. Θεωρούμε ότι τα κράτη-μέλη πρέπει να έχουν όσο το δυνατόν πιο ευρείες αιτίες, τις οποίες θα προβάλλουν για να αιτιολογήσουν σε περίπτωση που χρειαστεί να περάσουν στη φάση 2, σε περίπτωση που χρειαστεί λοιπόν να αιτιολογήσουν μια απαγορεύση. Αυτές είναι κύριε Πρόεδρε οι παρατηρήσεις μας για τα σημαντικότερα σημεία τα οποία έθιξαν τα μέλη της Επιτροπής σας εδώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον ε, Διευθυντή τον κύριο Πότλε και δίνω τώρα το λόγο στην κυρία Ρης για να κλείσει τη συζήτηση. Ευχαριστώ. Ε, εν συντομία θα μιλήσω. Δεν θα ξανανοίξω εδώ τη συζήτηση ολόκληρη. Αντιλαμβανόμαστε πόσο δύσκολη είναι η θέση η δική μου και όλων των συνεισηγητών, όλων των συνεισηγητών γενικά. Η κυρία Γιούσο και ένας ούγκρος συνάδελφος ε, είπαν την ουσία. Είναι θέμα ελευθερίας, την ελευθερία που πρέπει να διασφαλίσουμε και να παγιώσουμε για τα κράτη-μέλη που επιθυμούν να πούν όχι. Να συμφωνούμε από αυτού. Αλλά ανάλογα με το πώ θα εξηγήσουμε τα όσα μα προτείνει το Συμβούλιο, μπορεί να συμφωνούμε λιγότερο ή περισσότερο με τι προτάσει. Και αληθεύει ότι θα είναι δύσκολο ο συμβιβασμό. Εδώ αναφέρομαι στη φάση 1, η οποία σχολιάστηκε ευρέω και από μένα. Έχουμε τη θέση του κ. Στάση, τη κυρία Εβή, που λένε Όχι, δεν το θέλουμε, το απορρίπτουμε και άλλοι που θέλουν να διατηρηθεί. Θα είναι πολύ δύσκολο το να βρούμε συμβιβασμό για ζητήματα σαν αυτά. Θα ήθελα λοιπόν να κάνω μια πρόταση που αποσκοπεί σε δύο στόχους, διαφάνεια και αποτελεσματικότητα της διαδικασίας. Δεν είμαι βέβαιη, όπως λέει η Κομισιόν, η οποία φυσικά ναι, δεν επινόησε τη φάση 1. Δεν είμαι βέβαιος, βέβαιη ότι εδώ βρισκόμαστε σε απόλυτη ασφαλεία δικαίου. Άκουσα τις ερωτήσεις του Ζιλπαρνιού Ποιο σα εγγυάται ότι το κρατό ε, θα είναι σε θέση να μπορεί να προβάλλει όλε τι αιτιολογίε που ε, προτείνουμε να παρουσιάζει εδώ στη φάση 1. Εδώ έχουμε ένα δεσμευτικό κείμενο, έχουμε μια οδηγία και αυτή η φάση 1 είναι κάποιο είδου ε, διαδικασία ήπιου δικαίου που δεν είναι επαρκής και θεωρούμε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εδώ πρέπει να τροποποιήσει το κείμενο γιατί αυτό το κομμάτι δεν είναι δεσμευτικό για κανέναν. Να απαντήσω στον κύριο Στάς γιατί δεν ξέρω αν μήπω ε, δεν κατάλαβε καλά κάτι. Είπε, και δεν ξέρω αν το λέει στο Συμβουλίο σε μένα, είπε ότι ο κατάλογος των αιτίων και των κριτηρίων εδώ δεν ήταν επαρκή και γιατί δεν επανήλθαμε στα κριτήρια του Κοινοβουλίου. Μα αυτό έκανα. Ίσως δεν κατάλαβε καλά. Ουσιαστικά εγώ θέλω να επανέλθουμε σε αυτά που συζητήθηκαν εδώ, που απαιτήθηκαν εδώ, που προβλήθηκαν εδώ ως επιχειρήματα τα, οι αιτίε αυτέ, ε, όχι με την ίδια ερμηνεία όπω αυτή τη Κομισιόν, αυτά που επιθυμούσε το Κοινοβούλιο ήδη πριν από τρία χρόνια. Όσο είμαστε πιο ακριβείς και δώσουμε αδιάστατα επιχειρήματα νομικά στα κράτη-μέλη, ώστε να μπορούν να υπερασπιστούν σε περίπτωση προσφυγής. Σε περίπτωση που χρειαστεί να υπερασπίσουν τις ε, αποφάσεις τους να πούν όχι στα προϊόντα αυτά. Και ε, αυτό βασίζεται και στην εμπειρία των κρατών μελών που βρέθηκαν σε τέτοια θέση. Πρέπει τα επιχειρήματα να είναι όσο το δυνατόν πιο ακριβή. Καταλαβαίνω τόσο είπε και η Γκέρλινγκ για τη βάση. Το έχουμε συζητήσει και καταλαβαίνω ότι λέει. Το έχουμε συζητήσει και με τους κοιόδες. Η βάση είναι το ζήτημα εδώ. Είναι κάτι συμβολικό. Αντιλαμβάνομαι ότι το προβάλλουν ως red line, ως κόκκινη γραμμή ορισμένα κρατημέλη, ορισμένες ομάδες, οι νομικές υπηρεσίες ε, δεν έχουν καταλήξει ακόμη σε συμπέρασμα όσον αφορά το ζήτημα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ναι, επιθυμεί μια νομική βάση βασισμένη στο περιβάλλον. Εμείς ε, έχουμε την οδηγία του 2001, αλλά το 2003 η οδηγία αυτή του 2003 έχει τρεις ε, νομικές βάσεις, ε, γεωργίας, υγείας και εσωτερικής αγοράς, οπότε το ζήτημα παραμένει σε εκκρεμότητα. Αλλά πιστεύω ότι βοηθώ λίγο στη συνοχή προτείνοντα και έτσι απαντώ στην κυρία Γκέρλινγκ, η οποία μου λέει γιατί παίρνουμε αυτό που ήταν η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο σύνολο. Κοιτάξτε, παίρνουμε αυτά τα οποία σχεδόν ομόφωνα είχαν γίνει αποδεκτά και επεξεργαζόμαστε αυτά. Δεν είναι ότι σβήνουμε το παρελθόν. Εγώ πιστεύω πάντως ότι άκουσα ομοφωνία στο δύσκολο ζήτημα της συνύπαρξης. Όλοι συμφωνούμε από αυτού. Και συμφωνώ με τον Ούγκρο συναδέλφο, τον κύριο Αντιπρόεδρο, ότι θα πρέπει να είμαστε πιο ακριβείς σε αυτή την τροπολογία όσον αφορά τις ζώνες ανάσχησης, τη κριτήρια για να μπορέσουμε να λύσουμε αυτό το θέμα της συνύπαρξης. Αλλά είδα ότι υπάρχουν κάποια σημεία στα οποία διαφωνούμε, οπότε θα συνεχίσουμε την εργασία μας, τη συνεργασία μας. Να σας αφήσω κύριε Πρόεδρε να συνεχίσετε το χρονοδιάγραμμα, γιατί όπως είπαμε δεν έχουμε πολύ χρόνο. Ευχαριστώ πολύ τη συναδελφό την κυρία Ωραία, το χρονοδιάγραμμα λοιπόν προβλέπει εξαιρετικά στενά περιθώρια. Έχουμε προθεσμία τροπολογιών 15 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ. Ψηφοφορία για την εντολή στην Επιτροπή Περιβάλλοντος στις 5 Νοεμβρίου και ε, δεχόμενη ψήφο επιβεβαίωση τη συμφωνία σε περίπτωση που επιτευχθεί συμφωνία με το Συμβούλιο τον Ιανουάριο του 2015 και ψηφοφορία στην Ολομέλεια του Ιανουαρίου 2015 μπορούμε να θεωρήσουμε ότι έχουμε ολοκληρώσει το σημείο αυτό της ημερήσιας διάταξης και να περάσουμε στο άλλο σημείο της ημερήσιας διάταξης το οποίο αφορά τα νέα τρόφιμα, τα novel foods. Να κάνουμε μια μικρή σύνοψη, ανακεφαλαίωση, ελπίζοντας ότι ο συνάδελφος, ο ε, κύριος συζητητής θα έρθει εγκαίρω ώστε να μην χρειαστεί να δικαστηθεί από τη συνάδελφο κυρία Ντέρλεγκ. Όπως γνωρίζετε για η σύσταση αυτή, για τα, η ρύθμιση για ο κανονισμός για τα νέα τρόφιμα έχει παλιά ιστορία. Δεδομένου ότι η πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου παρουσιάστηκε ε, από την Κομισιόν 14 Ιανουαρίου 2008. Η νομοθετική συζήτηση Δήρξε πολύ χρόνο και η Επιτροπή της Συνδιαλλαγής δεν κατάφερε να επιτυχεί τελική συμφωνία στην τελευταία του συνάντηση της 28 Μαρτίου του 2011. Γι' αυτό το λόγο η πρόταση δεν υιοθετήθηκε και δεν έγινε νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σήμερα βρισκόμαστε ενώπιον μιας πρότασης αρκετά πιο περιορισμένης σε σχέση με την προηγούμενη. και θα χρειαστεί να εκφέρουμε γνώμη. Η πρόταση αυτή αντιγράφει ένα κομμάτι των συμπερασμάτων που της Επιτροπής Συνδιαλλαγής συμπεράσματα για τα οποία υπήρχε μια αρκετά εκτενής πλειοψηφία. Δίνω, τώρα το λόγο στην συναδελφό Γκέρλινγκ εκ μέρους του κυρίου Σίγητη και μετά θα αρχίσουμε το γύρο τραπέζι για να ακούσουμε τι απόψει των διαφόρων πολιτικών ομάδων. Παρακαλώ, κύριε Λίνγκ. Ε, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Γκέρλινγκ. Διαβάζω αυτά που έχει διαβιβάσει, να διαβιβάσει μάλλον δύο μου προς εσάς ο κύριος Νίκολσον. Οπότε δεν φταίω εγώ για ό,τι θα ακούσετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ αυτό το, το, το, εργαστήριο που έγινε την Τρίτη. Ήταν πάρα πολύ συνθετικό ότι ήρθαν όλοι και οι ηγητέ και συμμετέχουν στη συζήτηση. Και ε, ευτυχώ ελπίζω μάλλον ότι όλοι θα διαβάσετε πριν τη σημερινή συνεδρίαση την έκθεσή μου και τι νομίζω ότι θα μπορέσετε να συμβάλλετε σε αυτό στο οποίο θα καταλήξουν προσπάθειε όλων των εμπλεκομένων και αυτό το οποίο επιθυμούμε όλοι οι εμπλεκόμενοι. Δηλαδή να υπάρχει μια πιο ε, ταχεία διαδικασία για τα νέα τρόφιμα και όσον αφορά τι τρίτε χώρε επίση και τι σχετικέ αδειοδοτήσει. Πιστεύω ότι θα καλύψουμε αυτό που θέλουν οι καταναλωτέ, η βιομηχανία και οι σκιώδει ηγητέ. Έκανα ό,τι μπορούσα γι' αυτό και εγώ ήθελα να μιλήσω για, για τα θέματα τα οποία έχουν θέσει οι σκιώδει ηγητέ και πώ τροπολογίζουμε ότι καλύπτουν ο, ο ορισμός του τι θα πει νέο τρόφιμο, αυτό συνεχίζει και είναι ένα βασικό θέμα διαφωνίας και συζήτησης. Θεωρώ ότι θα πρέπει να βοηθήσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σαν τόσο έχει πει για τον ορισμό, σε σχέση με το τι κατανάλωση σε, ε, ε, σε μεγάλο βαθμό σημαίνει στην πράξη. Οπότε έχω τις πέντε και 14. Αυτές οι τροπολογίες που αφορούν το τι θα γίνει μέχρι ότου τεθεί σε ισχύ αυτή η νομοθεσία. Αυτό σημαίνει ότι η βιομηχανία και οι καταναλωτές θα μπορούν να κάνουν ε, επιλογή για το τι θα παράγουν ή τι θα τρώγουν Ο κύριος Ποκ ε, είπε κάτι σε σχέση με αυτό που λέει στο άρθρο 2 Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκεί που λέει για τα φαγητά ε, τα, τα τρόφιμα τέλο πάντων. Αυτό σημαίνει όμως ότι θα έχουμε μια άλλη διαδικασία λήψης ε, αδειοδότησης. Αν θέλουμε κάπως να τονώσουμε την καινοτομία, να έχουμε λιγότερη γραφειοκρατία, και ε, τότε θα ε, έπρεπε να έχουμε άλλη αιτήψη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εγώ υπέβαλα σχετικώς μια τροπολογία. Και ο Σπόκ και η κυρία Μπόρεν επίσης είπαν ότι δεν παραπέμπω στη μελέτη περιοδών πτώσεων της Κομισιόν, όμως έχω μια τροπολογία για τη δεύτερη του λίγη παράγραφου, ούτω ώστε να έχουμε υψηλό επίπεδο προστασίας ε, το υγεία των καταναλωτών και του περιβάλλοντος. Και αυτό αφορά και την πολιτική που ασκεί η Ευρωπαϊκή Ένωση για τα είδη διατροφής. Οπότε τελικά ο, όλος ο κόσμος θέλει να γίνει μια αναθεώρηση και του θέμα του ορισμού γιατί πολλοί εδώ και στην Επιτροπή Γεωργίας έχουν προβληματιστεί για τον κλονισμό ε, ότι αυτό θα πρέπει να ισχύσει ή να μην ισχύσει λένε για τα νέα ε, τρόφιμα θα ήθελα το θέμα του κλονισμού, τη κλωνοποίηση τέλο πάντων και των νέων τροφίμων να προχωρήσουν παράλληλα, να λάβουμε επίση υπόψη την προϊστορία που υπάρχει για αυτό το νομοθέτημα. Όλοι θέλουν κάποια ασφάλεια και βεβαιότητα. Ε, και επομένω δεν θα πρέπει να αποτελούν όμοιρου, επειδή το θέλουν αυτό οι, οι καταναλωτέ. Ε, οπότε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει κάνει το διαχωρισμό μεταξύ τη κλωνοποίηση και του νέου τροφίμου. Εγώ θα σα τονίσω ότι τα κλοπημένα τρόφιμα θα πρέπει να ρυθμιστούν χωριστά και γι' αυτό και δεν έχω απαλείψει τη μνήμα τη μέλου σα οδηγία από την έκθεση. Σύμφωνα με τον κύριο Στά, ότι θα πρέπει να υπάρχουν σωστά μεταβατικά μέτρα τα οποία να θεσμοθετηθούν και στι επαφέ μου και με την Επιτροπή αλλά και με το Συμβούλιο μου βεβαίωσαν ότι θα υπάρχει κάποιο είδου κενό στον νόμο εάν δεν περάσουν τα δύο σχετικά νομοθετήματα ταυτόχρονα. Και τώρα θέλω να στραφώ στο θέμα των νανοηλικών. Ε, τα νανοηλικά είναι ένα πάρα πολύ περιπλημμένο θέμα και οπότε θεώρησα ότι δεν πρέπει να κάνω τροποποίηση στην σχετική διάταξη για να διαφυλαχθεί η ασφαλεία δικαίου. Επίσης είμαι ανοιχτό στα επιχείρηματά σας. Στην τρίτη στο εργαστήρι είδαμε ότι τα νανοηλικά παραμένουν ένα θέμα επίμαχο για πολλούς. Επομένως, τι θα γίνει και πώς θα μπορούσαμε να τονώσουμε καινοτομία και επενδύσεις. Και αυτό το ποσοστό για το κατόφλι μπορεί να αποτελέσει φραγμό και τροχοπέδι. Τρόσον αφορά τις εφαρμοστικές πράξεις, τις πράξεις κατευθυνσιοδότηση. και εδώ έχουμε μια σειρά από επιχειρήματα και ξέρω ότι η Επιτροπή Εμπορίου και η Επιτροπή Γεωργίας θέλουν να αλλάξουμε ε, να γίνουν πράξη του ξεδότης και όχι εφαρμοστικέ. Οπότε έτσι να έχει το Κοινοβούλιο τον πρώτο λόγο, αλλά δεν ξέρω αν το Συμβούλιο θα το βρει εύκολο να συμφωνήσει. Κυρία Γιούσο, μας μίλησε για την προστασία των δεδομένων στο παρελθόν και νομίζω ότι συμφωνούμε και δύο ότι θέλουμε περισσότερη και λιγότερη συνεργασία μεταξύ επιστημόνων και βιομηχανία για την παραγωγή αυτών των καινοτόμων προϊόντων. Ελπίζω ότι η τροπολογία με υπαριθμών 24 θα το καταφέρει αυτό. Ο κύριο Στάς επίσης λέει ότι προβληματίζεται στον το θέμα της διαφάνειας. Εγώ είμαι υπέρ του να έχουμε πλήρη διαφάνεια και σε σχέση με αυτή την λίστα των νέων τροφίμων. Δεν μπορώ να σας... Ε, δεν έχω το χρόνο να σας ε, πω για τις άλλες τροπολογίες, αλλά σας είπα τα βασικά που με απασχολούν, εμένα, τους σκιώδες, την, κατά ε, τους καταναλωτές και τη βιομηχανία σε σχέση με την προτάσταση της Επιτροπής. Και όπως είπα και στο εργαστήρι. Ε, περιμένω να υποβάλλετε τις τροπολογίες σας τις αμέσως επόμενες ε, μέρες. Ελπίζω να έχουμε συνένεση και αυτός είναι ο σκοπός μου, ελπίζω να μαζί να το καταφέρουμε. Α, να και ο κύριος Νίκολσον και έχει τώρα τη σκητάλη. Ευχαριστώ, δεν ξέρω αν ο κύριος Νίκολσον θα ήθελε να προσθέσει κάτι. Όχι. Παρακαλώ. Ευχαριστώ την κυρία Γκέρλιν πάρα πολύ για τις παρατηρήσεις της, αλλά επειδή όλοι Δεν έχω ειδική τετριότητα και δεν μπορώ να σας βοηθήσω. Η κυρία Αγιούζο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πρώτα πρώτα να συγχαρώ τον κύριο Νίκολσον και την κυρία Γκέρλινγκ που τοποθετήθηκε αντί για εκείνον όσον αφορά αυτήν την ε, έκθεση η οποία πραγματικά καλύπτει όλες μου τις ανησυχίες σε σχέση με όλα όλα για την πρόταση της Επιτροπής. Πρώτα πρώτα για τις νέες κατηγορίες όσον αφορά τον ορισμό των νέων τροφίμων. Νομίζω ότι αυτό είναι το πιο καυτό θέμα. Α, αυτό ανησυχεί όλο τον κόσμο για αυτές τις κατηγορίες που υπήρχαν στον κανονισμό τον προηγούμενο του 1997 Ελπίζουμε ότι θα αποφύγουμε το να μην υπάρχει ασφαλεία δικαίου και να έχουμε επίσης σαφή ορισμό και να ξέρουμε τι είναι νέο και τι δεν είναι νέο τρόφιμο. Επίσης, τι αποτελεί παραδοσιακό προϊόν τρίτης χώρας ή τι είναι ασφαλής διατροφική χρήση κάποιου τροφίμου. Τώρα όσον αφορά τις προθεσμίες και εδώ σύμφωνα με τον εισηγητή ότι σε διάφορες φάσεις της διαδικασίας πρέπει να έχουμε ξεκάθαρες προθεσμίες. Έτσι κι αλλιώς. Θα πρέπει να δείξουμε ευελιξία. Και από την αποκεντρωμένη να πάμε σε μια συγκεντρωτική διαδικασία για την νέα διαδικασία αυτός ο μήνας για την υποβολή των στοιχείων ε, στην ΕΦΣΑ. Συμφωνώ ότι θα πρέπει να υπάρχει αυτή η τε, η τετράμινη για να υποβληθεί ε, αυτή η εκτελεστική πράξη στην ε, Επιτροπή, την αρμόδια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Να δούμε. Βέβαια, εάν είναι ρεαλιστικές οι προθεσμίες που προτείνει ο εισηγητής. Συμπαθάτε με τώρα όμως γιατί θα πρέπει να φύγω, γιατί πρέπει να πάω στην ε, συνεδρία της Επιτροπής με τις, για τις σχέσεις με την Χιλή. Ευχαριστούμε. Σωστή ομάδα, κύριο Πότσο. Ευχαριστώ. Συγχαρητήρια. Βελτιώνονται τις πρότασεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και η θέση του Συμβουλίου και το ότι ξαναμπαίνουν εδώ διαφορετικές κατηγορίες για τον ορισμό του νέου τροφίμου. Έχουμε επίσης και πνευματικές ρήτρες, κάπου νομίζω στην δεύτερη τροπολογία. Τώρα έχω και κάποιες παρατηρήσεις. Είχαμε προσπαθήσει να επικυροποιήσουμε την νομοθεσία και δεν καταφέραμε γιατί υπήρχαν ζητήματα κάποιων προϊόντων από κλωνοποιημένα ζώα κλπ. Τώρα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει η κλωνοποίηση να αποτελέσει αντικείμενο άλλης νομοθεσίας. Βέβαια, θα πρέπει να επιταχυνθούν οι διαπραγματεύσει και το νομοθέτημα που έτσι καλώς αρχίσει να συζητείτε να τεθεί σε ισχύ όσο γίνεται νωρίτερα με κάποια μεταβατικά μέτρα. Σας παραπέμπω τώρα στην τροπολογία 32 του εισηγητού. Επίσης, και το, η παραπομπή στην ε, ε θέση εμπορία προϊόντων που προέρχονται από ζώα, κάτι το οποίο ε, μας οδηγεί μετά αυτή την τροπολογία στο να διαγραφεί σχετική παράγραφος του άρθρου 1. Επίσης θα πρέπει στις ε, κατηγορίες που προτείνει εδώ η συγητής, θα πρέπει να παράγουμε και κάποιους ιστούς που προέρχονται από ζώα που μεγάλωσαν σε, σε πειραματικές. Πάντως είναι πρόβλημα και τα νανοηλικά. Λέει αναλυτικά ο σχετικός κανονισμός. Ο 1169 του 11 που αφορά την ενημέρωση του καταναλωτή για τα είδη διατροφής. Παίρνει θέμα εδώ για το θεσίες και λοιπά. Για το 50% των ανοηλικών είναι ένα κατόφλιο στον πρώτο χαρακτηρισμό. Δεν συμφωνεί εύσα πέραν αυτών των να έχουμε πάνω από 50% να νανοηλικά σε κάποια ιδιοτροφή. Επίση, μήπω μπορεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή ο εισηγητή να μα αναλύσουν λίγο περισσότερο τι γίνεται όσον αφορά την προστασία των δεδομένων στην τροπολογία 91 συγκεκριμένα λέει ότι θα υπάρξει προστασία δεδομένων όποτε έχουμε μελέτη επιστημονικού περιοδικού. Γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην αρχή είχε πει ότι θα έχουμε προστασία δεδομένων μόνο δεν έχουμε θέμα δημοσίευση. Κυρία Πόλσεν, ευχαριστώ, πρόεδρε. Να ευχαριστήσω ιδιαίτερα ε, την κυρία, τον κύριο Νίκολσον. Θεωρώ ότι η πρόταση είναι καλώς και πολύ σωστή. Είμαι ιδιαίτερο ικανοποιημένη για την ιδέα να επανέλθουν οι κατηγορίες, γιατί θεωρώ ότι γίνεται έτσι πιο συγκεκριμένη η πρόταση και μας διευκρινίζει καλύτερα τι είναι τα νέα τρόφιμα. Αυτό είναι σημαντικό, γιατί με πάσα ειλικρίνη η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ήταν μάλλον ασαφής. Εμείς λοιπόν θα υποστηρίξουμε ουσιαστικά όλες αυτές τις προτάσεις. Το μόνο που θα ήθελα να εξετάσουμε λίγο πιο προσεκτικά είναι το σημείο που αφορά την περιβαλλοντική αξιολόγηση των νέων προϊόντων. Προκειμένου να συμπεριληφθεί λοιπόν αυτό το στοιχείο, θα εξετάσω κατά πόσον υπάρχει χώρος στο κείμενο, στο διδακτικό δηλαδή του κειμένου, γιατί στην παρούσα φάση περιοριζόμαστε σε αναφορά στα... στις σκέψει. σκέψεις. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν αυτό. Θα πρέπει να αξιολογηθεί ο συνολικός κίνδυνος. Θα το εξετάσω και θα δω πώς μπορούμε να το εντάξουμε στο κείμενο, στο διδακτικό. Ευχαριστώ όμως και πάλι. Κύριε Νίκολσον, ήταν πραγματικά εξαιρετική πρόταση. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος, την κυρία Πόλσον και τώρα το λόγο έχει ε, ο συνάδελφος Μπόιλαν. Η συνάδελφος Μπόιλαν. Ευχαριστώ πρόεδρε. Να ευχαριστήσω τον εισηγητή για τη δουλειά που έχει κάνει μέχρι σήμερα για το θέμα αυτό. Παρ' όλα αυτά θα πρέπει να τονίσω κάποιες ανησυχίες που αφορούν διάφορες πτυχές της ε, πρότασης. Η, η καθυστέρηση για τις επιχειρήσεις μπορεί να αποτελέσει πολύ απογοητευτικό στοιχείο και γι' αυτό λοιπόν θέλω να μην υπάρχουν όπου είναι περιττές οι καθυστερήσεις. Αλλά μόνο όσο δεν υπάρχει κίνδυνο σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση κινδύνου των νέων τροφίμων. Είναι πάρα πολύ απαραίτητο λοιπόν να υπάρχει ε, η αρχή της αναλογικότητας. Ιδιαίτερα όταν μιλάμε για νέα τρόφιμα στην ευρωπαϊκή αγορά και γι' αυτό λοιπόν λυπάμαι που δεν αναφέρεται αυτή η βασική αρχή ούτε στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ούτε στο σχέδιο έκθεσης του εισηγητή. Επίσης πολύ λυπάμαι. Δεν θα ήθελα να υπάρξουν ε, προθεσμίες σε ό,τι αφορά προϊόντα που έχουν χρησιμοποιηθεί με και έχουν κατασκευαστεί με νανοτεχνολογία, γιατί δεν υπάρχει κάποιο ασφαλές επίπεδο νανοτεχνολογίας για το τρόφιμα και επίσης δεν υπάρχει οικονομικά βιώσιμος τρόπος να εξετάσουμε τα νανοελικά. Θα πρέπει λοιπόν να μην προτρέχουμε σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση τέτοιων νέων τροφίμων. Αν παραμείνουν οι κατηγορίες, πιο σωστό και πιο ασφαλές θεωρώ θα ήταν να μην επεξεργαζόμαστε, να μην μεταχειριζόμαστε τα τρόφιμα από τεχνολογία με τον ίδιο τρόπο ή σε ό,τι αφορά παράδειγμα τρόφιμα που παράγονται από μύκητες ή από φύκια. Είναι διαφορετικές οι κατηγορίες αυτές. Δεν θα πρέπει να επιτρέψουμε νέα τρόφιμα τα οποία δεν έχουν επιστημονική σφραγίδα να περνάνε γρήγορα γρήγορα. Θα ήθελα διευκρινήσεις επίσης σε ό,τι αφορά τα επιπρόσθετα στοιχεία της έκθεσης. Η έκθεση, όπως και η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αναφέρει ότι τα τρόφιμα από τρίτες χώρες που θεωρούνται νέα τρόφιμα θα πρέπει να θεωρούνται ασφαλή μόνο αν προέρχονται από την πρωτογενή παραγωγή όπως ορίζεται από τον κανονισμό 178 του 2002. Έχω μπροστά μου τον κανονισμό. Τι σημαίνει αυτή η πρωτογενή καταπαραγωγή. Πρωτογενή προϊόντα που συμπεριλαμβάνουν τη συγκομιδή, την, τα γαλακτοκομικά, την αλληλεία, το κυνήγι. Ουσιαστικά όλα λοιπόν τα τρόφιμα συμπεριλαμβάνονται. Δεν είναι λοιπόν λάθος να συμπεριλαμβάνονται όλα αυτά τα πρωτογενή τρόφιμα. Μήπως είναι υπερβολικά ευρύο το πεδίο εφαρμογής. Θα ήθελα λοιπόν μια διευκρίνηση και ιδιαίτερα όπως αναφέρεται στην ιδεολογική σκέψη 12 ανεξάρτητα αναφέρεται από τα αν είναι μεταποιημένα ή μη. Επιπλέον, επίσης, μια διευκρίνηση θα ήθελα για το πώς εννοείται τις νέες παραγωγικές διαδικασίες που μπορούν να ισχύουν για το τρόφιμα και τι χρονικό περιορισμών. Επίσης, τρόφιμα τα οποία προέρχονται από τέτοιες χώρε θα πρέπει να εκλέχονται πιο επισταμένος. Θα ήθελα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς την κατεύθυνση αυτή να κινηθεί. Ο Επίτροπος ο εισηγητής αναφέρει ότι αναφέρεται μάλλον η έκφραση αν είναι το τρόφιμο, αν δεν είναι σημαντικά λιγότερο θρεπτικό από το προηγούμενο τρόφιμο, σε σχέση με το προηγούμενο τρόφιμο. Ε, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σαφές αυτό και είναι νομικά αβέβαιο το τι εννοείται. Επίσης ε, για την αλλαγή της διατύπωσης σε ό,τι αφορά τον αντίκτυπο στην ανθρώπινη υγεία ε, αναφέρεται πλέον κίνδυνος για την υγεία και έτσι διευκρινίζεται πιο σωστά το τι ε, πρέπει να περιληφθεί. Και επειδή είναι δύσκολο ακόμα και να εντοπιστούν τα νονό ε, στοιχεία στο τρόφιμα. Καλό είναι λοιπόν να περιορίσουμε το πεδίο εφαρμογή. Και τέλο, επειδή μιλάμε για, το, τρόφιμα και για τη δημόσια υγεία, η παρακολούθηση μετά το μάρκετινγκ θα πρέπει να αποτελεί τον κανόνα για όλα τα τρόφιμα και όχι κάτι προαιρετικό ή ε, σε περιπτώσεις που δικαιολογείται μόνο όπως αναφέρει ο εισηγητής. Άρα προσβλέπω στη συνεργασία με τους κοιότης για να βελτιωθεί περαιτέρω το κείμενο αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Το λόγο έχει ο συνάδελφος ο κ. Στάες. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εφτά σημεία έχω να θέξω. Πρώτον, το ανέφερε και η κυρία Μπόιλαν. Η αρχή της ε, πρόληψης. Πολύ βασικό στοιχείο για όλη την ομοθεσία. Τη στηρίζω. Να κάνουμε μια κοινή τραπολογία. Δεύτερο στοιχείο. Αυτό που δεν ε, συμπεριλαμβάνεται στην όλη ιστορία σήμερα είναι που τα νέα τρόφιμα αποφέρουν ωφέλη καινούργια για τους καταναλωτές. Θεωρώ ότι αν πρέπει να υπάρχει ένα νέο τρόφιμο θα πρέπει να υπάρχει και κάποιο όφελος για τον καταναλωτή και θα πρέπει να προσταθεί αυτό ως διάσταση. Τρίτο, τι κάνουμε με τα τρόφιμα από ζώα. Στο κείμενο της κυρίας Γκέρλινγκ που είχε κατακτήσει ο εισηγητής αναφέρεται ότι η νομική βεβαιότητα μετά από μια μεταβατική περίοδο και ότι υπήρξαν επαφές με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θεωρώ ότι θα πρέπει να το σκεφτούμε αυτό. Εμάς μας ανησυχεί ως πράσινους, γιατί δεν θέλουμε να υπάρχουν νομικά κενά. Θέλουμε να φροντίσουμε η νομοθεσία για τα νέα τρόφιμα να φροντίσει να ξέρουμε καλά τι γίνεται ανα πάσα στιγμή και πότε θα τεθούν σε εφαρμογή οι νομοθεσίε που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θεωρώ ότι αυτό εκ παραλίλου θα πρέπει να τεθεί σε εφαρμογή. Τέταρτο στοιχείο. Νάνο τεχνολογία. Ο κύριο Πόκ το ανέφερε. Εργαζόμαστε αυτή τη στιγμή με τον ορισμό που βρίσκεται υπό αναθεώρηση. Υποβάλαμε και μια ένσταση σε ό,τι αφορά την νομοθεσία για την ε, πληροφόρηση των καταναλωτών για τα τρόφιμα. Εδώ χρησιμοποιούμε το όριο του 50%, αλλά όντως αυτό ισχύει για την επισήμανση. Εδώ μιλάμε για άλλο κινδύνου. Η ΕΦΣΑ όμως, η αρχή ασφάλειας των τροφίμων, συστήνει να εφαρμόσουμε ένα κατόφλι 10%. Θεωρώ ότι είναι ένα στοιχείο αυτό. Δεν πρόκειται να αγγίξουμε την νομοθεσία για την επισήμανση. Βλέπω ο κόσμος με κοιτάει με τρόμο. Αλλά εδώ, σε αυτόν τον ορισμό, θεωρώ ότι θα έπρεπε να μπορούμε να το συζητήσουμε το θέμα αυτό. Και θεωρώ ότι είναι συντηρητική η προσέγγιση μας. Ε, καλύτερα να ακολουθήσουμε την πρόταση του 10% της ΕΨΑ. Πέμπτο. Η όλη συζήτηση για τις πράξεις κατά εξουσιοδότηση, τις εφαρμοστικές πράξεις, ο εισηγητής λέει ότι θα είναι δύσκολες οι συζητήσεις με το Συμβούλιο, δεν θέλει να ακούσει τίποτα το Συμβούλιο, αλλά θεωρώ ότι θα πρέπει να τηρήσουμε θέση αμετακίνητη ως Κοινοβούλιο. Γιατί να μην χρησιμοποιήσουμε τις πράξεις κατά εξουσιοδότηση για τέτοια ζητήματα. Αν ξέρουμε για παράδειγμα ότι τα νέα τρόφιμα με τις εφαρμοστικές πράξεις θα μπορούσαν να εγκριθούν χωρίς να μην υπάρχει οποιαδήποτε περιθώριο να πει τη γνώμη του το Κοινοβούλιο. Ενώ άλλα ισχύουν για τα πρόσθετα των τροφίμων, τα χρωστικά, που είναι η λογική. Γιατί το ένα να το κάνουμε με πράξη κατεξουσιοδότησης και το άλλο όχι θεωρώ ότι θα πρέπει να τα δώσουμε τον αγώνα αυτό. Το πρώτο τελευταίο σημείο τώρα, το έκτο σημείο, η συμμετοχή της ΕΦΣΑ. Τώρα το άρθρο 9.2 αναφέρει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενδέχεται, may, να ζητήσει την ε, έγκριση της ΕΦΣΑ. Εδώ θεωρώ ότι θα πρέπει να επανέλθουμε στην προηγούμενη πρόταση, όπου ήταν σαφές ότι η ΕΦΣΑ πάντα θα πρέπει να γνωμοδοτεί. Και τέλος, τελευταίο σημείο σε ό,τι αφορά την διαφάνεια. Το είχα αναφέρει και στην αρχή στον εισηγητή, στον κ. Νίκολσον και χαίρομαι ιδιαιτέρως για την αντίδρασή του, το ότι έχει δείξει ανοιχτό πνεύμα. Σίγουρα θα καταθέσουμε σχετικέ τροπολογίες και ελπίζω να καταλήξουμε σε μια συμφωνία για το θέμα αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Τελευταίος ομιλητής, η συνάδελφος κυρία Εύη, εξ των ομάδων. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, το ζήτημα του ορισμού των novel food ε, για μας δεν πρέπει να περιορίσουμε το πεδίο του ορισμού, διότι θεωρούμε ότι βρισκόμαστε ενώπιον ε, ενός ε, τομέα που εξελίσσεται διαρκώς. Δεν μπορούμε να τον προβλέψουμε. Το να προσπαθήσουμε να τον ορίσουμε υπερβολικά επακριβώς μπορεί να αποδειχθεί αντιπαραγωγικό. Όσον αφορά όμω τα παραδοσιακά τρόφιμα, Δηλαδή τον αυτοματισμό που αναφέρεται στο κείμενο μπορεί να μην προστατεύει απόλυτα έναν πληθυσμό που πάει να χρησιμοποιήσει νέα υλικά τα οποία δεν έχει συνηθίσει. Ε, κάποια παραδοσιακά τρόφιμα ορισμένων πληθυσμών μπορεί να αποτελέσουν πρόβλημα για άλλους πληθυσμούς. Ε, Λείπουν λοιπόν κάποιες προϋποθέσεις για να μπορέσει να οριστεί το επίπεδο ασφαλείας επειδή δεν υπάρχουν επαρκείς επιδημιολογικές μελέτες. Ένα παράδειγμα, σαφές, είναι η δυσανεξία στην ε, γλουτένη λόγω ειδών σιτηρών που αναπτύχθηκαν με την πρώτη γεωργική επανάσταση αλλά για την οποία δεν υπάρχουν επιδημιολογικές μελέτες. Ε, συνεπώς δεν συμφωνούμε με τα όσα αναφέρονται. Επίσης θεωρούμε ότι την κατάσταση ρουστροφίμου με ένα άλλο μπορεί να γίνει αποδεκτή εφόσον δεν υπάρχει μείζον κίνδυνο. Και αυτό είναι άλλο ένα στοιχείο το οποίο πρέπει να ληφθεί υπόψη. Η δυνατότητα να ορίσουμε ένα τρόφιμα είναι ή όχι νέο τρόφιμο πρέπει να ανατεθεί στην Κομισιόν, η οποία θα πρέπει να ζητήσει τη γνώμη της ΕΦΣΑ και όχι τα κράτη-μέλη αυτό ώστε να υπάρχει πιο ομοιόμορφη εφαρμογή του προτύπου στο κοινωτικό επίπεδο. Κάτι άλλο που προσδιορίσαμε τα κριτήρια αξιολόγησης των νέων τροφίμων πρέπει να μπορούν να συμπεριλάβουν το life cycle assessment, την αξιολόγηση κύκλου ζωής. Πέραν των διατροφικών χαρακτηριστικών πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και τις κοινωνικές επιπτώσεις αυτών των νέων τροφίμων. άλλα δύο σημεία που έχουμε εντοπίσει. Το άρθρο 22. Η προστασία δεν μπορεί να καλύπτει τις απαγορεύσεις ε, της πληροφορίας υγείας δηλαδή και η πρόταση τροποποίησης του άρθρου 23 ε, δεν μας βρίσκει σύμφωνος. Η τροπολογία 88 που σχετίζεται με το άρθρο 23 αντιθέτως αφορά τις πληροφορίες ασφαλείας δεν μπορούν να καλύπτονται από βιομηχανικό απόρριτο και αυτό είναι κάτι που θέλουμε να υπογραμμιστεί. Και τέλος, όσον αφορά το ποσοστό νανοηλικών, θεωρούμε και εμείς ότι η ένδειξη του 10% της ΕΦΣΑ πρέπει να ληφθεί υπόψη. Οποιοδήποτε μεγαλύτερο ποσοστό, οτιδήποτε έχει μεγαλύτερο ποσοστό θα θεωρείται ότι είναι novel food. Ευχαριστώ. ευχαριστώ. Ας περάσουμε στις άλλες παρεμβάσεις των συναδέλφων. Παρακαλώ περιοριστείτε στα τρία λεπτά το πολύ, ώστε να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε έγκαιρα. Θα ξεκινήσω με τη συνάδελφο Σέγια Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σε ό,τι αφορά τις προτάσεις του εισηγητή, σε ό,τι αφορά τη συζήτηση για τα τρόφιμα, θα πρέπει να μην ξεχνάμε ότι τα νέα τρόφιμα είναι μια νέα ευκαιρία, αν θέλουμε να συνεχίσουμε να έχουμε τρόφιμα για όλο τον κόσμο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν αυτό να υπάρχει και μια κοινωτική προσέγγιση. Θα πρέπει να μην υπάρχει κατακαιρματισμό. Σε ό,τι αφορά τον ορισμό, θα πρέπει να φροντίσουμε να μην υπάρχουν εξαντλητικοί κατάλογοι. Θα πρέπει να έχουν ευελιξία τα κράτη-μέλη προκειμένου να θεωρούν ως ε, νέα τρόφιμα τα κράτη-μέλη, αν το επιθυμούν. Και τέλος, θα πρέπει πρωτογενής, πρώτη ευθύνη να είναι αυτή του παραγωγού, για να αποφασίζει και να είναι υπεύθυνος για το αν είναι νέο τρόφιμο ή όχι, το τρόφιμο που παραγάγει. Και αυτό την προηγούμενη εβδομάδα συζητήθηκε και θα πρέπει να έχουμε υπόψη ότι πρόκειται για το περιβάλλον, για την δημόσια υγεία, αλλά το πιο βασικό είναι η ασφάλεια των τροφίμων για όλη την, ε, για όλη εφήλιο. Ευχαριστώ, συνάδελφος Καπούτο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι πολύ σύντομος, επειδή πολλά ήδη υπόθηκαν. Ήθελα να κάνω κάποιες διευκρινήσεις. Πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τον κύριο Σιγητή ο οποίος ε, επανησύγαγε την κατηγορία των novel food που την είχαμε ξεχάσει. Πέραν της ασφάλειας δικαίου, αυτή η κατηγορία εφαρμόζεται σε ορισμένα προϊόντα μόνο. Υπάρχει το θέμα της κλωνοποίησης που πολλοί ανέφεραν ήδη. Εδώ η Ευρωπαϊκή Ένωση πληρώνει το τίμημα του νομοθετικού κενού που έχει ε, πιστεύω ότι πρέπει να επικεντρωθούμε σε μεταβατικά μέτρα τα οποία θα επιτρέψουν την εφαρμογή του κανονισμού για τα νέα τρόφιμα όσον αφορά τα προϊόντα που προέρχονται από κλωνοποιημένα ζώα μόνο εφόσον έχει διευκρινιστεί η έγκριση της νέας οδηγίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η το ζήτημα των κατεξοδότηση πράξεων. Εδώ φυσικά εμείς ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να κάνουμε μια προσπάθεια να αποκτάμε όλο και περισσότερες εξουσίες. Ε, θεωρώ ότι είναι σημαντικό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να έχει τη δυνατότητα να ελέγξει τους καταλόγους προϊόντων καθώς ε, εμπλουτίζονται αυτές οι καταλογοί. Όσον αφορά τις νανοτεχνολογίες, ο συνάδελφος Πόσα ήδη είπε, ανέφερε τη θέση της ομάδας μας. Θεωρώ ότι πρέπει να συμφωνήσουμε στο μέγιστο δυνατό βαθμό με τη θέση της ΕΦΣΑ γιατί πρέπει να εγγυηθούμε την ασφάλεια των καταναλωτών κυρίως. Υπάρχει ένας ορισμός ε, που δεν έχει αναλυθεί επαρκώς σε σημαντικό ποσοστό που βρίσκεται, χαρακτηρίζει το κείμενο και θα πρέπει να διευκρινιστεί. Πρέπει δηλαδή να ορίσουμε παραμέτρους αναφοράς ε, αρκετά αντικειμενικές. Θεμελιώδη ρόλο θα πρέπει να διαδραματίσει φυσικά η ΕΦΣΑ, ενδεχομένως σε συντονισμό με τα κράτη-μέλη και με τη Συμβουλευτική Επιτροπή για τα Νέα Τρόφιμα που υπάρχει ήδη. Τέλος, μια τελευταία σκέψη για τα παραδοσιακά ε, τρόφιμα από τρίτες χώρες. Εγώ θα πρότεινα και εδώ εφόσον δεν υπάρξουν αιτιολογημένες αντιρρήσεις, να περνούν αυτόματα από μια πλήρη αξιολόγηση κινδύνου στην ΕΦΣΑ, στην αρχή της διαδικασίας. Ευχαριστούμε. Το λόγο έχει η συνάλφωση κυρία Γκαρντίνη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι και εγώ σύντομη. Χαιρετίζω το γεγονός ότι εδώ περιοριζόμαστε στην ασφάλεια των νέων διατροφικών προϊόντων και αφήνουμε στο πλάι όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με την κλεονοποίηση των ζώων, με των ε, εκτρεφόμενων ζώων, διότι εγώ ήμουν μέλος της ε, αντιπροσωπείας ε, που είχε πάει για διαπραγματεύσεις και θυμάμαι πώς έγινε εκείνη η διαπραγμάτευση. Και είμαι βέβαιη ότι θα ξαναβρεθούμε σε αδιέξοδο, να πρέπει ξανά δηλαδή τα νέα τρόφιμα να τα βάλουμε στην άκρη. Διότι γνωρίζουμε τις θέσεις που έχουν διατυπωθεί. Χαιρετίζω λοιπόν αυτή την επιλογή, αλλά θεωρώ ότι έχει γίνει μεγάλο κομμάτι της δουλειάς ήδη. Εδώ είναι έτοιμο, διότι υπήρχε αρκετά ευρεία συμφωνία. Παρότι ο τομέας αυτός είναι τόσο ευαίσθητος, εγώ θα ήθελα να κάνω μια πρόταση, δεν ξέρω αν μπορείτε να δεχτείτε χωρίς να επηρεαστούν το συνολικό χρονοδιάγραμμα, διότι όλοι θέλουμε φυσικά η εργασία αυτή να ολοκληρωθεί κατά το Ιταλικό εξάμεινο. Αλλά, δεδομένου ότι αύριο θα συνεδριάσει μια ομάδα εργασίας στο Συμβούλιο ε, για τα νέα τρόφιμα Αντί η προθεσμία για τις τροπολογίες να είναι η Παρασκευή, δεν θα μπορούσαμε να έχουμε κάνα δύο μέρες παραπάνω, γιατί κοιτάξτε, εδώ έχουμε ένα ζήτημα τόσο ευαίσθητο που για να σταθμίσουμε σωστά τις διάφορες, τα διάφορα συμπεράσματα αυτής της ομάδας εργασίας και να μην κάνουμε λάθη, γιατί το θέμα αυτό είναι τόσο ευαίσθητο που αν δεν το ρυθμίσουμε καλά μπορεί να έχει σημαντικές επιπτώσεις 24-48 ώρες παραπάνω δεν αλλάζει πολλά πράγματα ε, ε, γενικώ, αλλά θα μας επιτρέψει να εμβαθύνουμε λιγάκι. Ζητάω πραγματικά, κάνω έκκληση, αν είναι δυνατόν, καλό θα ήταν, για να μην ε, βάλουμε λάθος πράγματα, να προλάβουμε να τα σκεφτούμε όλα καλά και να ξέρουμε τι κάνουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Και τώρα ο συνάδελφος κύριος Μπάτσο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Γνωρίζω καλά και κατάλαβα καλά ότι φτάνουμε στο τέλος μιας μακράς νομοθετικής διαδικασίας και τώρα πρέπει να το κλείσουμε. Αλλά θα ήθελα να σας πω την άποψή μου ως Ευρωβουλευτής. Μας είπαν ότι αυτή η πρόταση πρέπει να σέβεται την αρχή της επικουρικότητας και μετά είπαμε ότι τα κράτη-μέλη δεν μπορούν από μόνα τους ε, να επιτύχουν τους στόχους αυτής της πρότασης. Γιατί, διότι τα κράτη-μέλη με τις επιμέρους διαδικασίες τους θα ε, επιτύχαν ένα κατακαιρματισμένο ε, επίπεδο ασφάλειας ενώ χρειάζεται ενωσιακή προσέγγιση. Εγώ πιστεύω ότι αυτή η προσέγγιση είναι λάθος. Σε πολλά κράτη-μέλη έχουμε μέτρα ασφαλείας και κριτήρια ασφαλείας πιο αυστηρά από αυτά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πιστεύω λοιπόν ότι ούτε εδώ έχουμε μια οδηγία, μια πρόταση. Έχουμε ένα κανονισμό. Έχουμε την ελεύθερη κυκλοφορία των τροφίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε ορισμένα κράτη-μέλη. Έχουμε κριτήρια ασφαλείας σε σχέση με αυτά τα τρόφιμα. Ε, η Κομισιόν λοιπόν προβάλλει την ελεύθερη κυκλοφορία των τροφίμων με το σχέδιό της. Πρέπει να δεχτούμε δηλαδή τα κριτήρια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θεωρώ λοιπόν ότι το κείμενο έπρεπε να είναι λιγότερο δεσμευτικό για να ορίσουμε αυτά τα κριτήρια σε κλίμακα Ευρωπαϊκή Ένωση, Αλλά η Κομισιόν προτείνει ένα κανονισμό, γεγονός που δίνει προτεραιότητα στην ελεύθερη κυκλοφορία, όπως είπα, και δεν επιτρέπει στα κράτη-μέλη να λάβουν τις δικές τους αποφάσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Να δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να μας εξηγήσει τη θέση τους. Merci beaucoup, Monsieur le Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να συνοψίσω σε έξι σημεία τις παρεμβάσεις των συναδέλφων σας. Το πρώτο αφορά την κλωνοποίηση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παράλληλα με την πρόταση για τα νέα τρόφιμα έκανε αυτή την πρόταση το τέλη του 2013 ώστε το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο φυσικά να μπορέσουν να συζητήσουν αυτές τις δύο προτάσεις μείζωνος σημασίας όπως υπενθυμίσαμε φυσικά το εκλογοποίηση είναι ένα σχέδιο κειμένου το οποίο δεν θα αφήσει αδιαφορό το Συμβούλιο ούτε το Κοινοβούλιο. Ωστόσο θα επιθυμούσαμε, επειδή θεωρούμε ότι η κλωνοποίηση ε, προκαλεί περισσότερες αντιμαχιες από τα νέα τρόφιμα, οι εξελίξει των συζητήσεων για τα νέα τρόφιμα λοιπόν θα επιθυμούσαμε να προχωρήσουν πιο γρήγορα διότι εκεί φυσικά υπάρχει και το θέμα τη καινοτομία για τι μικρομεσαίε επιχειρήσει. Σημαντικό θέμα. Ορισμένοι όμω από εσά ε, εκφράσετε την επιθυμία στο μεσοδιάστημα, δηλαδή πριν εγκριθεί και υιοθετηθεί το κείμενο για την κλωνοποίηση, η κατάσταση που αφορά τα τρόφιμα αποκλωνοποιημένα ζώα να έχει διευκρινιστεί. Για μας είναι σαφές ότι εφόσον δεν υπάρχει νέο κείμενο για την κλωνοποίηση, τα τρόφιμα βάσει ε, υλικών προερχόντων από κλωνοποιημένα ζώα, κρέας, γάλα, θα παραμείνουν ε, στην κατηγορία των νέων τροφίμων. Και συνεπώς, ε, αν υπάρχει κάποιο έτοιμα, παρότι δεν υπήρξε μέχρι στιγμής, ε, παρότι υπάρξει έτοιμα συγκεκριμένο, σε περίπτωση που υπάρχει έτοιμα συγκεκριμένο, θα αποτρέψει το αντικείμενο εξέταση από την ΕΦΣΑ. Όπω γνωρίζετε, στη μελλοντική πρόταση προβλέπεται τα τρόφιμα αυτά από κλωνοποιημένα ζώα να απογορευτούν. Αλλά θεωρούμε ότι στο μεσοδιάστημα χρειάζεται να υπάρχει μια καθαρή κατάσταση. Το δεύτερο σημείο αφορά τις, τους πιο σαφείς ορισμούς των υπολείπων νέων τροφίμων, εκτός των κλωνοποιημένων. Προφανώς ε, οτιδήποτε μπορεί να προσφέρει η νομική σαφήνεια ε, είναι φυσικά ευπρόσδεκτο, αλλά δεν πρέπει να είναι πολύ περιοριστικό. Έχουμε ένα κατάλογο προϊόντων, τα οποία μπορούν να κατηγοριοποιηθούν ως νέα τρόφιμα, βάσει του παλιού κανονισμού, και είχαμε προβλήματα, για παράδειγμα, κατάταξης των εντόμων. Ένα σκορπιός ε, είναι νέο τρόφιμο ή όχι. Οποιοςδήποτε λοιπόν πολύ περιοριστικός ορισμός μπορεί να οδηγήσει σε νομική ασάφεια. Είμαστε σίγουρα λοιπόν υπέρ σαφών ορισμών φυσικά. Γι' αυτό που είμαστε πιο διστακτικοί είναι το τρίτο σημείο, τη πιο σύντομε προθεσμίε. Αντιλαμβανόμαστε ότι η βιομηχανία χρειάζεται σύντομε προθεσμίε ώστε να μπορέσει να έχει πολύ γρήγορα την άδεια κυκλοφορία στην αγορά ενό νέου τροφίμου. Αλλά Έχουμε διοικητικέ διαδικασίε, διυπηρεσιακέ διαβουλεύσει, μεταφράσει ε, και ούτω καθεξής. Σε επίπεδο κομισιών ε, δεν επιθυμούμε οι προθεσμίες να είναι πολύ σύντομε, οι οποίες αντίθετα με ότι ε, θεωρούσαμε μπορεί να μην με επιτρέψουν να εξετάσουμε ικανοποιητικά το θέμα. Το τέταρτο επιχείρημα αφορά τις νανοτεχνολογίες. Η ΕΦΣΑ μιλά για 10% στην επιστημονική της νομοδότηση. Αλλά σήμερα, όπως και οι Αμερικανοί και οι Καναδοί και οι Αυστραλοί φίλοι μας, βρισκόμαστε ενώπιον της αδυναμίας διαγνωστικού ελέγχου ενός ε, συστατικού, εάν περιέχει κάτω από 50% νανοσωματίδια. Το 10% από διαγνωστική άποψη δεν είναι εφικτό σήμερα και μας λυπεί αυτό διότι θεωρούμε ότι σε θέματα νεοτροφίμων το κατόφλιο του 10% για την επισήμανση ειδικότερα είναι αναγκαίο κατόφλιο αλλά όσο οι εργαστηριακές τεχνικές δεν είναι σε θέση να προσδιορίσουν αν ε, το ποσοστό είναι 10, 20, 30, 40% νανοσωματιδίων σε ένα συστατικό θεωρούμε ότι δεν μας ικανοποιεί να αναφέρεται αυτό το κατόφλιο. Αντιθέτω, ε, στη μελλοντική κατεξοδότηση πράξη που συζητάμε αυτή τη στιγμή, θεωρούμε ότι το κατόφλιο αυτό που σήμερα είναι 50% θα μπορούσε να αναθεωρηθεί σε συνάρτηση με τις εργαστηριακές τεχνικές. Μόλις οι τεχνικοί εμπειρογνώμονες και αυτό επιβεβαιωθεί από την ΕΦΣΑ μας πούν ότι μπορούμε να κάνουμε διάγνωση με βεβαιότητα και χωρίς ε, ε, αμφιβολία ποσοστά 10, 20, 30% τότε δεσμευόμαστε να περάσουμε σε αυτό το χαμηλότερο κατόφλιο, διότι αντιλαμβανόμαστε πολύ καλά τις ανησυχίες των καταναλωτών και την επιθυμία τους να ενημερώνονται. Και ότι ε, το να γνωρίζει κανείς ε, το 10, 20, 30% διασφαλίζει τη ασφαλειά του. Το κατόφλιο αυτό είναι κατόφλιο που θα αναφέρεται στην επισήμαση δεν είναι κατόφλιο ασφαλείας. Το πέμπτο σημείο αφορά την προστασία των δεδομένων. Θεωρούμε ότι πρέπει να ευθυγραμμίζεται με τον κανονισμό που αφορά τους ισχυρισμού, τα claims. Θεωρούμε ότι δεν πρέπει να υπάρχει διαφορά, διότι αυτό θα ήταν επιζήμιο για τις βιομηχανίες, ε, να υπάρχουν δύο νομοθεσίες διαφορετικού τύπου. Φυσικά χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Αφενός Πρέπει να προστατεύσουμε την καινοτομία και τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας. Αφετέρου, πρέπει οι επιχειρήσεις να έχουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν και αυτές νέα προϊόντα. Θεωρούμε λοιπόν εμείς ότι σκόπιμο είναι να είμαστε προσεκτικοί. Τέλος θα ολοκληρώσω με τις κατεξουδότηση πράξεις. Οι κατεξουδότηση πράξεις και όπως γνωρίζετε στην ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή που έρχεται, όταν θέσετε εγκρίνει όλους τους ε, επιτρόπους, προβλέπετε ότι το Κοινοβούλιο θα εμπλέκεται πολύ περισσότερο, ειδικότερα στην εκπόνηση των της πράξεων. Και θα μπορείτε, όπως ήδη τώρα, αλλά ίσως πιο συστηματικά στο μέλλον, θα μπορείτε να προβλέψετε μεγαλύτερη συμμετοχή του προσωπικού του Κοινοβουλίου στην προετοιμασία των κατεξίδων αυτών αυτών από την Κομισιόν. Γεγονός που θα σας επιτρέψει σε πρώιμο στάδιο να γνωρίζετε τις προθέσεις της Επιτροπής. Θα σας δίνει επίσης περισσότερες δυνατότητες αντίδρασης σε περίπτωση που υπάρχουν προτάσεις κατεξοδότηση πράξεων που δεν σας βρίσκουν σύμφωνος. Τέλος κύριε Πρόεδρε για να ολοκληρώσω θα ήθελα να πω ότι εμείς συνεργαζόμαστε στενά με τον εισηγητή τον κύριο Νίκολσον και τους Σκιώδης ώστε αυτή η έκθεση και οι συζητήσεις σας να μπορέσουν να προχωρήσουν πολύ γρήγορα με ελπίζουμε συμφωνία με το Συμβούλιο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε την Κομισιόν και για τις τεχνικές πληροφορίες που μας παρήχε να δώσω το λόγο στον κύριο Νίκολσον για να κλείσει τη συζήτηση. Ε, thank you very much. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ Πρόεδρε και επειδή έχει περάσει και η ώρα θα είμαι πάρα πολύ σύντομος. Ε, όπως όλοι ξέρουμε είναι πολύ τεχνικής φύσεως η εκθεσία αυτή και ξέρω ότι κάποιοι συνάδελφοι έθεσαν κάποια ερωτήματα σήμερα και καλύτερα κάποια από τα ζητήματα αυτά να συζητηθούν σε επίπεδο μεταξύ των ειδικών για τα νοηλικά, για παράδειγμα. Αυτό σίγουρα θα μας απασχολήσει ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τα θέματα συναπόφασης προκειμένου να υπενθυμίσω στην Επιτροπή ότι οι εμπειρογνώμονες στο Συμβούλιο ούτε αυτοί μπορούν να συμφωνήσουν μεταξύ τους. Αυτό είναι μάλλον ενθαρρυντικό. Θα πρέπει λοιπόν να πετύχουμε κάτι σωστό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό όπως τόνισαν και διάφοροι συνάδελφοι. Υπάρχουν και κάποια άλλα θέματα. Ρωτήσατε για το κατά πόσο θα μπορούσε να παραταθεί. Εγώ από τους άλλους εξαρτάμαι. Εγώ θα ήθελα να παρατείνω τη διαδικασία, αλλά εξαρτάμαι από τη γραμματεία. Αν οι τροπολογίες παραταθούν μέχρι τη Δευτέρα, όλοι ταξιδεύουν και πήγαινε στο Στρασβούργο, δεν ξέρω κατά πόσο θα βολεύει αυτό. Θα χάναμε χρόνο δηλαδή ουσιαστικά. Και δεν θα είχαμε τη μετάφραση στη τελική ανάλυση. Γνέψτε κατεφαντικά, αν δίκιο έχω. Ναι, δεν προλαβαίνουμε τη μετάφραση για την ε, ψηφοφορία τη Δευτέρα στο Στρασβούργο το Νοέμβριο. Αν λοιπόν μπορείτε να το αποδεχτείτε αυτό, εγώ ναι, ευχαρίστω να έδινα πιο πολύ χρόνο. Αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση νομίζω πιο σημαντικό είναι να μπορέσουμε να ψηφίσουμε στο Στρασβούργο. Κατανόηση λοιπόν ζητώ. Και ίσω να πρέπει αυτή την εβδομάδα να δουλέψουμε λίγο πιο σκληρά. Κατά τα άλλα θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφου και όλε τις ε, άλλε παρεμβάσει. Ε, και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και προσβλέπω στη συνεργασία με τους Κιώδης. Στο μέλλον θεωρώ ότι θα πετύχουμε καλά αποτελέσματα μόλις λάβουμε και τις τροπολογίες να δούμε πού μπορούμε να φτιάξουμε συμβαστικές τροπολογίες. Ευχαριστώ Πρόεδρα. Ευχαριστούμε James. Και τώρα το χρονοδιάγραμμα. Όπως είπατε θα ήταν πολύ δύσκολο να έχουμε τη μεταφράση των τροπολογιών έγκαιρα για τις επόμενες συνεδριάσεις, διότι την, η επόμενη εβδομάδα είναι εβδομάδα Στρασβούργου. Και στο Στρασβούργο δυστυχώς ε, θα είναι πολύ πιο δύσκολο να τα κλείσουμε όλα για να τα στείλουμε για μετάφραση. Παραμένουμε λοιπόν με το χρονοδιάγραμμα που είχαμε προβλέψει με προθεσμία για τις τροπολογίες 17 Οκτωβρίου 10 το πρωί. Η επόμενη συνεδρία της Επιτροπής ε, για την ε, μελέτη των τροπολογιών 5-6 ε, Νοεμβρίου. Ψηφοφορία στην Επιτροπή ΕΜΒΗ σε μια έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής μας 24 Νοεμβρίου στο Στρασβούργο. έχουμε φτάσει στο σημείο που έχουμε κλείσει τα σημεία της ημερησίας διάταξης ε, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σας ευχαριστώ για τη συμμετοχή σας στη συνεδρίασή μας και μπορούμε να θεωρήσουμε ότι έχει κλείσει η συνεδρίαση της Επιτροπής και περνάμε στη συνεδρία των συντονιστών. Parlamentar